good afternoon, ladies and gentlemen, and um, welcome to um, our. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζουμε σήμερα και αύριο πρωί και απόγευμα. Τελευταία φορά πριν από τα τέλη Αυγούστου που θα ξανασυνεδριάσουμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν όλοι. Ε, υπάρχει αναμετάδοση μέσω του διαδικτύου της συνεδρίασης αυτής να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, παρακαλώ. Η κυρία Στήλερ όμως έχει κάτι να πει. Ε? Να... Πρέπει να φύγετε, οπότε θέλετε πιο γρήγορα να εξετάσουμε το δικό σας θέμα. Ναι. Να δούμε. Θα δείτε επίσης το IMCO News. Ε? Πίσω στην αίθουσα υπάρχουν αντίγραφα και στα έδρανα. Επίσης να σας πω ότι αύριο το πρωί, όχι αύριο το απόγευμα, θα συναντηθούμε με τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, τον Πολωνό, αύριο. Να είσαστε εδώ λοιπόν, παρακαλώ, αύριο το απόγευμα για την συνάντηση αυτή. Έχουμε και ένα μήνυμα από την Προεδρία που είναι κάτι που έχουμε προσθέσει στο έγγραφο εδώ, στο IMCO News. Για τα πρακτικά τώρα, της 24ης και 25ης Μαΐου. Υπάρχουν τα πρακτικά στους φακέλους σας. Αν δεν εκφράσετε κάποια αντίρρηση, κάποιο σχόλιο μέχρι τη λήξη της συνεδρίασής μας αύριο το βράδυ, θεωρούνται εγκεκριμένα. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, να συνεχίσουμε και περνάμε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Πρόκειται για τον εξυγχρονισμό της πολιτικής δημόσιων συμβάσεων. Όπως ξέρετε, Πολλοί από εσά είχαμε ήδη μια κρόση και τώρα έχουμε ένα σχέδιο έκθεση τη συζητήτριά μα, τη κυρία Ρούλε, η οποία θα μα παρουσιάσει και το θέμα αυτό. Μετά θα ακούσουμε του σκιώδει συζητητέ, τον κύριο Ένβα από το ΕΛΚΑ, την κυρία Βανιού από του Σοσιαλιστέ, τον κύριο Κρόιτσμαν από την Άλντε και εγώ θα παρέμβω από το ΙΣΙΑΡ. Ο κύριος Δεγιόγκ δεν είναι εδώ, ούτε κανένα άλλος. Αυτά από τους Σκιώδης. Και μετά η κυρία Στερ Σμιτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάρει το λόγο, η οποία θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Χωρίς άλλη καθυστέρηση, λοιπόν, δίνω το λόγο στην Χάιντι Ρούλε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω δύο παρατηρήσεις τεχνικής ε, φύσεως. Θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω, αν θέλετε να δουλέψετε με την ε, γερμανική εκδοχή, να προσέξετε λιγάκι ε, το νόημα ε, γιατί υπήρχε μεγάλη πίεση χρόνου. Ε, την Παρασκευή το μεσημέρι συνέταξα τις τροπολογίες και ε, όταν επρόκειτο να ε, επανεπεξεργαστούμε τα 21 άρθρα είπαμε ότι καλύτερα να τα συντάξουμε από την αρχή. Τώρα λοιπόν υπάρχει στο διαδίκτυο η σωστή διατύπωση. Θα δω λιγάκι και πώς ε, είναι η διατύπωση στα γαλλικά. Πάντως να σας πω στο πρώτο κομμάτι η πρωτότυπη διατύπωση είναι στα γερμανικά και μετά στα αγγλικά. Και το έκανα αυτό συνειδητά. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Η δεύτερη μου παρατήρηση είναι η εξή. Για όσου θέλουν να καταθέσουν τροπολογίε, θα ήθελα να σα παρακαλέσω να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με του σκιώδει ηγητέ και του έχω ήδη δώσει τι δικέ μου τι ε, τροπολογίε. Βεβαίω, 6.000 ε, ε, στοιχεία είναι πάρα πολλά αν θέλει κανείς να έχει δύο πράσινες βίβλους. Στο δεύτερο τμήμα αναγκάστηκα να προσθέσω κάποιες παραγράφους που δεν υπήρχαν στο πρώτο. Ε, Παραδείγματος χάρη και που γίνεται λόγο για τη διαφθορά, ε, για την χρηστή διαχείριση. Ε, αυτά προσθέτηκαν και ως έκτο κομμάτι όλο αυτό που αφορά την ε, ηλεκτρονική ανάθεση έργων και από πλευρά ε, περιεχομένου θέλω να σας πω ότι τώρα πλέον είμαι σαφέστερη στο σχέδιό μου γιατί είχα περισσότερο χώρο και γιατί εντωμεταξύ έλαβα και τις ε, τροπολογίες, τις αλλαγέ τη ε, Κομισιόν. Αυτό για μένα που είναι πολύ σημαντικό και αναφέρεται στην, στο επεξηγηματικό σημείωμα είναι ότι ειδικά στον τομέα των δημόσιων διαγωνισμών χρειαζόμαστε το διάλογο ανάμεσα στους αναθέτοντες και ανάμεσα στους ιδιώτες ε, μειοδότες, γιατί για τους δεύτερους ισχύει θα πρέπει να έχουν γνώσεις της αγοράς, να εξοικειωθούν με ένα προϊόν ε, πριν συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό. Ε, στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει κάποια σάφια, πολλοί πιστεύουν ότι δεν επιτρέπεται πριν από τους διαγωνισμούς να κάνουν έρευνες αγοράς και φοβούνται ότι θα έχουν νομικές συνέπειες. Γι' αυτό για μένα το θέμα της πρόσβασης στην αγορά, ο διάλογος ανάμεσα στο δημόσιο και την αγορά θα πρέπει να εξαστεί καλύτερα. Και αυτό και έγινε. Κατόπιν ε, στις ε, τροπολογίες ε, εξετάζουν και αυτό το κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό και οδηγεί σε πολλές συζητήσεις στις οριακές τιμές. Στις ε, τιμές κατόφλι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη τιμή, κατά πόσον αυτέ τι τιμέ ε, κατόφλι θα πρέπει να τι αυξήσουμε ή όχι. Και αυτά στηρίζονται με αριθμού που αναφέρονται στη μελέτη τη Επιτροπή, ότι δηλαδή μόνο 1,6% ε, των αναθέσεων έργων ε, γίνεται διασυνοριακά. Όσον αφορά τώρα τις ε, τιμές, μιλάμε για 3,5% του όγκου, ε, μιλάμε για πολύ χαμηλές ε, τιμές και αν αυτά τα συγκρίνει κανείς με το ότι ένας δημόσιος διαγωνισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη στοιχίζει επιπρόσθετα 25.000 ευρώ, πολλοί μειοδότες που βρίσκονται κυρίως στο κατώτερο κομμάτι διορωτώνται γιατί θα πρέπει οι διαγωνισμοί να γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει. Ε, Βεβαίω, εγώ τώρα δεν δεσμεύομαι, αλλά καλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μα δώσει περισσότερε πληροφορίε επί του θέματο, ε, διότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αρκετέ συγκεκριμένε πληροφορίε για το θέμα. Και το, οι μικρομεσαίες επιχειρήσει και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να επεξεργαστούμε. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα όπου υπάρχουν ασάφειες Πρόκειται για τους ε, περίφημους ε, κοινούς διαγωνισμούς ε, και τις ομάδες συμμετεχόντων. Στην Ευρώπη Υπάρχει το εξή θέμα. Πολλοί φοβούνται ότι η διαγωνίτα γίνεται μόνο μία φορά το χρόνο και πολλές μικρές επιχειρήσεις φοβούνται ότι αν συγκεντρώνονται πολλές επιχειρήσεις αυτές θα ζημιωθούν. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι όσον αφορά τις κοινού τους κοινούς δημόσιους διαγωνισμούς και την ομαδοποίηση των προσφορών. Εκεί η Γερμανία είναι πολύ πιο προχωρημένη από άλλε χώρε. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι ακριβώ προτείνουν. Εγώ δεν έχω ακόμα διαμορφώσει άποψη και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφή η διατύπωση. Κατόπιν ε, και το θέμα των προδιαγραφών και αυτό κατά την άποψή μου δεν περιλαμβάνεται όμως το θέμα των προδιαγραφών ε, το συζητήσαμε στην τελευταία μου έκθεση πέρυσι γι' αυτό σε αυτή την έκθεση είμαι λίγο πιο σύντομη επί του θέματος ε, και αν θέλετε να έχετε και τις ε, δύο εκθέσεις και τη δεύτερη που περιλαμβάνονται οι τροπολογίες μου ευχαρίστω να σας τις στείλω για να δείτε τι έχει προσθεθεί επιπρόσθετα στην έκθεσή μου νομίζω το σημαντικότερο μήνυμα είναι εκείνο το οποίο κατέστη σαφέ στη διάσκεψη των Προέδρων αλλά και σε όλες τις ε, τοποθετήσεις για την Πράσινη Βίβλο. Χρειαζόμαστε λοιπόν απλούστευση των ε, κανονισμών για τους δημόσιους διαγωνισμούς, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία και σε ορισμένου τομεί ε, χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη νομική σαφήνεια, σαφής, σαφέστερη διατύπωση. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα επιτύχουμε το δεύτερο στόχο μας που είναι εξίσου σημαντικός, δηλαδή η ανάθεση έργων, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο όπου διερχόμαστε οικονομική κρίση, τέτοιου είδους αναθέσεις, αυτή την περίοδο πρέπει να τύχουν ε, σωστής εκμετάλλευσης, Μιλάει πάρα πολύ γρήγορα η ομιλήτρια, ε, υπερβολικά γρήγορα και ο πρόεδρος του διακόπτη. Επαναλαμβάνει λοιπόν η ομιλήτρια. Για μένα είναι σημαντικό να γίνεται στρατηγική χρήση της δημόσιας ανάθεσης έργων έτσι ώστε σε περίοδους κρίσης οι αναθέσεις έργων αποτελούν ναύσματα για καινοτομίες, για ε, βιώσιμη ανάπτυξη και για συνοχή. Το σημαντικότερο σημείο, ε, το σημαντικότερο μέσο με το οποίο μπορεί κανείς να τα επιτύχει όλα αυτά είναι η απλούστευση των κανονισμών και η μεγαλύτερη ευελιξία. Παράλληλα όμως υπάρχουν και εργαλεία ε, τα οποία οι αναθέτοντες ε, πρέπει να τα χρησιμοποιούν σωστά και ο καθένας να γνωρίζει τι μπορεί να χρησιμοποιήσει. Υπάρχει το θέμα των διαδικασιών διαπραγματεύσεων και βεβαίως ε, στις διαπραγματεύσεις να υπάρχουν και τα απαραίτητα εχέγγυα, διαφάνεια και ούτω καθεξής. Υπάρχει και το θέμα της χρήσης ε, εναλλακτικών λύσεων, εναλλακτικών προτάσεων που και αυτές πρέπει να ενισχυθούν. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές δυνατότητες και τέλος Θέλω να θίξω ένα θέμα ε, για το οποίο επίσης πρέπει να συζητήσουμε. Κατά την άποψή μου, η ερμηνεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο του, ε, σχετικά με τα τεύχη δημοπράτησης ε, είναι πολύ περιοριστική η ερμηνεία αυτή. Ε, καταρχήν γίνεται λόγο, ή γίνεται αναφορά αν θέλετε στο προϊόν και όχι στη μέθοδο παραγωγής. Αν όμω θέλουμε να προάγουμε καινοτόμα προϊόντα ή την ε, βιώσιμη ανάπτυξη αυτό που παίζει ρόλο κατά κύριο λόγο είναι η μέθοδος παραγωγής. Γιατί σε ένα καινοτόμο προϊόν μπορεί κανείς να δει πώς έχει παραχθεί. Παραδείγματο χάρη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτές παράγονται με διαφορετικό τρόπο από τις συμβατικές μορφές. Αυτό όμως δεν το βλέπουμε στο τελικό προϊόν, μόνο στη μέθοδο παραγωγής. Και το ίδιο συμβαίνει και σε άλλους τομείς. Παραδείγματο χάρη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Σουηδία τρεις ε, δίκες ε, που ε, τρέχουν. Πρόκειται για το catering, ε, για τα ζωικά προϊόντα και για τον τρόπο εκτροφής ζώων. Εγώ θέλω να πω ότι η μέθοδο παραγωγή πρέπει να λαμβάνεται εξίσου υπόψη όπω και το προϊόν. Από την άλλη επιθυμώ να υπάρχει και μία διευκρίνηση. Δηλαδή να μην αναφέρεται ότι η αναφορά στο αντικείμενο θα πρέπει να αποδυναμωθεί. Γιατί πιστεύω ότι η σαφή αναφορά στο αντικείμενο του διαγωνισμού είναι πολύ σημαντική αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και τη δωροδοκία. Ε, και γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει αυτό το εχέγγυο. Και φτάνω στην τελευταία μου παρατήρηση. Όπως σας είπα, ε, συμπεριλαμβάνω στην έκθεσή μου και το θέμα της διαφθοράς. Ε, πιστεύω όμως ότι στη διαφθορά υπάρχουν ήδη σαφείς κανονισμοί. Και όσον αφορά το dumping, προσφορές dumping, το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού, εγώ με πέρα του να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Μόνο ε, που πρέπει αυτοί να είναι σαφείς για όσους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε μιλήσει για πολύ καιρό στην Πολωνία το να κατακυρωθεί ένας διαγωνισμός ε, στην Κίνα αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευθεί εάν είχαν αποκλειστεί οι τιμές dumping αν αυτό ήταν ευθύ εξ αρχής σαφές γιατί το προϊόν των Κινέζων ήταν κατά το ίμιση φθηνότερο από αυτό που υπολόγιζε η πολωνική κυβέρνηση. Ήταν ένα προϊόν κατά πολύ κάτω από την τιμή των προϊόντων που προσφέρονται στην αγορά. Ε, κατά την άποψή μου λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να ε, δημιουργήσουμε, να εφεύρουμε εμεί επιπρόσθετα εργαλεία, απλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά που υπάρχουν, να υπάρχει σωστή ενημέρωση και σωστή χρήση των ήδη υφιστάμενων εργαλείων και μέσων. Α, ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν τη σαφέστατη παρουσίαση. Τώρα θα μιλήσουν οι σκιώδεις και μετά όποιος άλλος θέλει να λάβει το λόγο. Ο κύριος Έγκελ. Κύριε Πρόεδρε, η παρουσίαση αυτή βασίζεται στο ίδιο πνεύμα με την περσινή μας εξέταση ενός παρόμοιου θέματος και γι' αυτό μπορούμε να παρακολουθήσουμε εύκολα αυτά που μας είπε. Και είναι επίσης εύκολο να γνωρίζουμε όλοι ποιες είναι οι βάσεις της μελλοντικής της τελικής έκθεσης. Αυτές οι βάσεις λοιπόν είναι η απλοποίηση, η νομική ασφάλεια και, και οι ή τα προμήθειες έτσι το λέμε στα γαλλικά, ή procurement. Όπως είπα λοιπόν και πέρυσι περίπου αυτά συζητήσαμε, τρία όμως θέματα θέλω να σχολιάσω με ορισμένες τροπολογίες. Μετά από αυτά που είπαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο, βέβαια είναι πιο εύκολη η συνένεση. Πρώτον, για τις υπηρεσίες και πέρυσι το είχαμε συζητήσει. Συνεχίζω να πιστεύω ότι ακόμη κι αν ορισμένοι στην Κομισιόν υπάλληλοι, όχι επίτροποι, μερικοί μουστερίδες στην Κομισιόν θέλουν να παραβιάσουν την περσινή συμφωνία δεν έχουν αποδείξει ότι υπάρχουν διαστρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς. Γι' αυτό θα θέλαμε όπως και πέρυσι να μάθουμε για ποιους λόγους αυτοί οι υπάλληλοι της Κομισιόν θέλουν να, οπωσδήποτε να μας επιβάλλουν πρόσθετη νομοθεσία για τις υπηρεσίες, κάτι για το οποίο το Κοινοβούλιο έχει εκφραστεί και άλλη φορά εναντίον. Για τα κριτήρια της οικονομικότερης προσφοράς τώρα. Συμφωνώ με τη σκέψη της κυρίας Ρούλε, αλλά ως προς τη διατύπωση θα μπορούσαν να υπάρξουν βελτιώσεις. Γιατί δεν καταλαβαίνω Πώς θα μπορούσε ο Ευρωπαίος νομοθέτης, όχι για αυτή την έκθεση αλλά για άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσε να μην εφαρμόσει αυτή την αρχή της οικονομικότερης προσφοράς, της φτηνότερης προσφοράς. Αν θέλουμε να την αντικαταστήσουμε με, να αντικαταστήσουμε τη φτηνότερη προσφορά με την οικονομικό συμφερότερη νομίζουμε ότι θα ήταν μια βελτίωση. Τέλος για τη διαφθορά. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και σε αυτό το επίπεδο των προσφορών και των ε, προμηθειών το να υποκρινόμαστε ότι, ότι μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις μεταξύ των τομέων ως προς τη διαφθορά νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα θα δούμε πως θα το διατυπώσουμε δεν είμαι κατά των διαπραγματευομένων αγορών αλλά αλλά διαφορά μπορεί να υπάρχει παντού. Τέλος. Κανονικά θα έπρεπε να προσθέσω και άλλα σχόλια για τον, την ηλεκτρονοποίηση των δημοσίων αγορών αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή και ελπίζω τελικά να υπάρξει συνένεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ συγχαίρω την Χάιντε για το κείμενό της που ευθυγραμμίζεται, όπως είπε και ο κύριος Έγγελς, τα όσα συμφωνήσαμε εδώ και έχουμε συζητήσει εδώ από πέρυσι. Δεν υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις. Η έκθεση ευθυγραμμίζεται απόλυτα στους άξονες που κατά προτεραιότητα επιθυμούμε εμείς και που περιλαμβάνονται στην πρόταση της Κομισιόν, δηλαδή απλοποίηση, που είναι κάτι αναγκαίο, και, όπως είπε και η συγκήτρια, χρήση των δημοσίων αγορών υπέρ των τομεακών πολιτικών στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Και αυτήν πρέπει να έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας. Συμφωνώ με τον κύριο Χέγγελ για αυτά που είπε για τα δέκα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί η σωστή διατύπωση. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να λέμε ότι η πιο φτηνή προσφορά είναι και η καλύτερη πάντα. Νομίζω ότι διατυπώνεται καλά. Μπορεί να βελτιωθεί ακόμα η διατύπωση. Η πιο ευνοϊκή οικονομικά προσφορά. Ναι, μην ξεχνάμε ότι αν δεν πάρουμε την πιο φτηνή λύση πρέπει πάντα να δικαιολογούμε γιατί. Αλλιώ ο κανόνας είναι η πιο φτηνή προσφορά. Λοιπόν, όντως είμαστε πολύ κοντά στην σωστή διατύπωση. Άρα εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Έρχομαι τώρα σε κάτι άλλο που η ομάδα μου, οι σοσιαλιστές, πιστεύει ότι μπορεί να βελτιωθεί. Το είπα και σε μια προηγούμενη συνεδρίαση. Δηλαδή, οι κοινωνικές πτυχές στις συμβάσεις, στις δημόσιες. Όταν έχουμε δηλαδή ξένες επιχειρήσεις για παράδειγμα που έρχονται και οι οποίες δεν συμμορφώνονται απαραίτητα με το δικό μας το δίκαιο όπως το υπενθυμίζουμε και το έχουμε υπενθυμίσει πρόσφατα στο κείμενό μας για την εσωτερική αγορά. Πρόκειται για τα δικαιώματα των εργαζομένων στις δημόσιες συμβάσεις. Είναι μικρές οι μεσές επιχειρήσεις που παίρνουν υπεργολαβία. Εδώ λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε πολύ καλά ποια είναι τα δικαιώματα και κυρίως ποιες είναι οι υποχρεώσεις αυτών των επιχειρήσεων που δρούν υπεργολαβικά, αλλά και των επιχειρήσεων εκείνων που χρησιμοποιούν τις πιο μικρές αυτές επιχειρήσεις υπεργολαβικά. Κατά τα άλλα, το είπε και η Χάιντε, τα θεμελιώδη είναι πολύ... Ε, βασικά και μας βρίσκουν σύμφωνος, υπάρχει το παράδειγμα αυτό της Πολωνίας με την Κίνα Ίσως θα πρέπει εδώ να προσθέσουμε και άλλα πιο συγκεκριμένα κριτήρια για τις συμβάσεις που κάνουμε με χώρες εκτός Ευρώπης. Υπάρχει και κάτι άλλο που θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε, το είπε λίγο και η Χάιντι. Όταν αναφερθήκατε στις μεθόδους παραγωγής, είδα τι λέτε για το fair trade, για το σωστό το δίκαιο εμπόριο. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και κάτι για τα κριτήρια που διέπουν το εμπόριο αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους πολίτες αλλά και για το περιβάλλον, όπως επίσης και για τις κοινωνικές πτυχές. Ένα άλλο σημείο το οποίο μας ανέφεραν μικρές επιχειρήσεις όταν πρόκειται για την πρόσβαση στις δημόσιες συμβάσεις. Και αυτό είναι η προστασία της καινοτομίας στα πλαίσια των δημοσίων συμβάσεων, όπου είναι υποψήφιες μικρές επιχειρήσεις. Φυσικά και πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, σχεδιασμός κτλ. Αλλά πρέπει να υπάρχει και το απόρριτο για να προστατεύονται οι μικρές αυτές επιχειρήσεις όταν καινοτομούν, γιατί είναι πολύ βασικό αυτό για την ανταγωνιστικότητά τους. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλα προβλήματα. Αλλά απ' την άλλη δεν συμφωνώ, βέβαια το λέω εκ μέρους μου και ίσως να συμφωνούν και μερικοί από την ομάδα μου για το εξή. Πιστεύω ότι όσον αφορά τα δικαιώματα τα δικαιώματα παραχώρησης, εδώ πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διευκρίνηση στην νομοθεσία. Υπάρχουν χώρες όπως η Πολωνία και άλλες που μόλις μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που ακόμα δεν έχουν μια αρκετά προχωρημένη νομοθεσία στον τομέα αυτό, το, στον τομέα των παραχωρήσεων. Υπάρχει ο κίνδυνος λοιπόν να υπάρξουν καταχρήσεις σε ορισμένες χώρες. Καλό θα ήταν η Επιτροπή να προσθέσει κάτι από αυτού. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι Ό,τι τροπολογίες υπάρχουν θα τις συζητήσουμε με την Χάιντι και θα δούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κρόιτσμαν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πραγματικά συγχαίρω την κυρία Ρούλε ε, για την πολύ καλή έκθεση και για την πολύ καλή ιδιαίτερα αγαστή συνεργασία που είχαμε. Όσον αφορά την ε, ανάθεση έργων. Ε, πράγματι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα. Οι οδηγίες ε, εγκρίθηκαν το 2004 και από την εμπειρία μου ξέρω πολύ καλά ότι χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο μέχρι να προσαρμοστούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να βιαστούμε ιδιαίτερα. Συμφωνώ ότι οι πανευρωπαϊκές ε, διαδικασίες ανάθεσης ε, έργων θα πρέπει να απλουστευτούν. Οι ηλεκτρονικές διαδικασίες ε, παίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά και η ίδια η οδηγία περί ανάθεσης δημόσιων έργων και αυτή θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Οι αρχές της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης, του θεμητού ανταγωνισμού, αυτές οι αρχές πρέπει να διατηρηθούν. Βεβαίως και η νομική έτσι ώστε ο τομέας εφαρμογής να μην περιορίζεται ε, κυρίως ε, να μην ε, προκύπτει αθέμητο όφελος. Τα κριτήρια θα πρέπει να ορίζονται σωστά. Επίσης είναι ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι οι δημόσιοι διαγωνισμοί μπορούν ε, να συμβάλλουν και στην επίτευξη πολιτικών στόχων. Η αρχή της εφαρμογής ε, του της οικονομικά ευνοϊκότερης ε, προσφοράς είναι σωστός δρόμος. Στη Γερμανία γνωρίζουμε ότι αυτή η αρχή πρέπει να διέπει την οικονομία. Η κυρία Ρούλε στην τηλεδιάσκεψη επισήμανε και το βρίσκω αυτό σημαντικό ότι μπορούμε να αποκλείσουμε την φτηνότερη προσφορά μέσα από την σωστή διατύπωση προδιαγραφών. Στους δημόσιους διαγωνισμούς θα πρέπει να προσέχουμε έτσι ώστε να υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες και όπου είναι σαφές είτε πρόκειται για βιβλία, αγορά βιβλίων είτε για χαρτί εκεί δεν πρόκειται και δεν είναι το σημαντικότερο η ευνοϊκότερη προσφορά έχω όμως ε, κατά νου τουλάχιστον από την εμπειρία μου ότι όταν εμείς ε, είχαμε δημοσιοι αγωνισμους ε, για αυτούς που φτιάχνουν τις στέγες εκεί οποτεδήποτε επιλέγαμε τον φτηνότερο έπεφτε η στέγη Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η δική μας εμπειρία στη Ρινανία Παλατινάτο και γι' αυτό λέμε ότι καλύτερα να πάρουμε όχι τους φτηνότερους αλλά τους ντόπιου ε, για να μπορούν μετά αν χρειαστεί να επισκευάσουν τη στέγη. Αυτή λοιπόν τη δυνατότητα πρέπει να την έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό υπάρχει στη Γερμανία. Δεν έχει νόημα να έχουμε πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς. Εξάλλου ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το σύνολο του κόστους. Αυτή η αρχή της ε, ευνοϊκότερης ε, προσφοράς δεν θα πρέπει να προβλέπει ότι επιλέγουμε το φτηνότερο προϊόν. Ισχύουν ε, κάποιες ε, δυνατότητες, κάποιες ε, προδιαγραφές Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθούμε να καλύπτουμε τα κριτήρια με κάποια αντικειμενικότητα. Διότι αλλιώς ε, καταλαβαίνετε ότι ανοίγουμε διάπλατα την πόρτα στην ε, διαφθορά και αυτό δεν το επιθυμούμε. Ίσως σε κάποιες ε, χώρες να είναι τα πράγματα καλύτερα από τις άλλες Όμω, ε, εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει περιττό γραφειοκρατικό κόστος και νομίζω ότι επίση αυτό που επιθυμεί η συνάρφωση η κυρία Ρούλε είναι το εξή όταν κάνουμε μία προσφορά θα πρέπει να υπάρχει έρευνα της αγοράς για να είναι η καλύτερη προσφορά. Και θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είναι πολύ ενδιαφέρον. Εμείς ε, κάποτε ε, είχαμε κάνει δημόσιο διαγωνισμό για την επισκευή αγωγών στο κανάλι που ήταν ακριβώς δίπλα από τα σπίτια. Ε, κάποια άλλη εταιρεία είπε αυτούς τους αγωγούς να τους βάλουμε στη μέση του ποταμού και να είναι πιο φτηνά. Μόνο που αυτή βέβαια ήταν κάποια ιδέα που άλλαζε τελείως τα πράγματα. Όταν λέμε ότι μιλάμε με την αγορά και με τους συμμετέχοντες στην αγορά, η ιδέα που θα επικρατήσει ενδεχομένως θα πρέπει να κοινοποιηθεί σε όλους εγώ σε επίπεδο αρχή συμφωνώ μαζί σα γιατί θέλω να πω ότι πράγματι ε, πρέπει να βρίσκουμε την φτηνότερη προσφορά όμως ε, η προσφορά θα πρέπει να είναι και καλύτερη να μην υπάρχει κανένα ίχνος ε, απάτης ε, στην όλη διαδικασία γιατί μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί. Η ιδέα είναι σωστή, κυρία Ρούλη την στηρίζουμε μόνο που πρέπει να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε και τι δρόμο θα βρούμε γιατί και οι ιδιώτες το κάνουν αυτό, εξετάζουν την αγορά και προσπαθούν να παρουσιάσουν την ευνοϊκότερη προσφορά. Συμφωνούμε λοιπόν με την ιδέα της ευνοϊκότερης ε, προσφοράς, μόνο που δεν έχουμε βρει ακόμα τη λύση για να μπορούμε να ε, συμπεριλάβουμε και την ε, προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Και κάτι άλλο, το οποίο αναφέρατε προηγουμένως. Διαπιστώσαμε στους δημόσιους διαγωνισμούς ότι οι πανευρωπαϊκοί διαγωνισμοί ίσως να είναι πιο δαπανηροί, αλλά από εκεί προκύπτουν οι ευνοϊκότερες τιμές. Γι' αυτό εγώ δεν θέλω να αλλάξει το θέμα των πανευρωπαϊκών διαγωνισμών. Κάνατε όμως μια πολύ καλή πρόταση. Πρέπει να δούμε τι συνέπειες για να το συζητήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ είμαι σκιώδης. Θα μιλήσω λοιπόν και εγώ. Θέλω απλώς να συμφωνήσω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε την Χάιντι για την εξαιρετική της έκθεση. Θα έλεγα ότι δύο είναι τα σχόλιά μου. Πρώτον είναι εξελικτική έκθεση γιατί σε σύγκριση με πέρυσι βλέπουμε πολλά κοινά στοιχεία. Η ανάλυση που έκανε η Επιτροπή μας δείχνει ότι η ανταπόκριση από την Κομισιόν με βάση το ερωτηματολόγιο της δείχνει ότι υπάρχει αρκετή ευθυγράμμιση μεταξύ των προβλημάτων που ταύτισε πέρυσι η κυρία Ρούλε στην Επιτροπή μας και το επιτροπή της Κομισιόν. Δεύτερον, θα έλεγα ότι η προσοχή που έδωσαν όλοι στην απλοποίηση της διαδικασίας χωρίς να απολεσθεί νομική ασφάλεια βεβαιότητα της διαδικασίας είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή λιγότερη γραφειοκρατία είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να είναι σαφές ότι πρέπει η διαδικασία να είναι ανταγωνιστική και ανοιχτή. Και επίσης σε σημαντικούς τομείς όπως τα πράσινα κριτήρια προμηθειών ή πράσινες παραγωγικές μεθόδους, όλα αυτά πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. Από το διαγωνισμό ήδη να τονίζεται αυτό. Να συνδυαστούν όλα αυτά λοιπόν, αυτό είναι η μεγάλη σημασία που έχει αυτή η έκθεση. Δεύτερον, ίσως λίγο πιο αμφιλεγόμενο, ότι η λογική της απλοποίησης των διαδικασιών αφορά τα κατώτατα όρια, τα κατόφλια, διότι το κόστος της προετοιμασίας διαγωνισμών συγκρινόμενο με την αξία του διαγωνισμού αυτού δεν είναι πάντα θετικό αν το κόστος, το κόστος δηλαδή μπορεί να είναι απαγορευτικό σε σύγκριση με τα ωφέλη. Τώρα βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα ως προς τα εργαλεία και την τεχνολογία που υπάρχει για τις δημόσιες προμήθειες. Πρέπει λοιπόν να ξαναπούμε ότι ακόμα και διαγωνισμοί που δεν ακολουθούν την πλήρη διαδικασία παρόλα αυτά πρέπει να συμφωνούν με ορισμένες ελάχιστες αρχές όπως την ίση μεταχείριση και τη διαφάνεια. Τώρα που πολλές δημόσιες αρχές χρησιμοποιούν το ίντερνετ για να δημοσιεύσουν διαγωνισμούς ή ακόμη και στην επίσημη εφημερίδα, μου φαίνεται ότι θα ήταν δυνατόν να καθοριστεί ένα συμβιβασμός μεταξύ της αύξησης των κατοφλίων και παράλληλα της σύνδεσης των στοιχείων αυτών με, τα Ευρωπα... με τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες Δεδομένων για λιγότερο σημαντικούς διαγωνισμούς που να συμπεριλαμβάνουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να διστάσουμε να το θίξουμε και αυτό. Ξέρω ότι τώρα θα διαφωνήσουν πολλοί, αλλά επειδή έχω ζητήσει καινοτομίε στον τομέα των δημοσίων προσφορών θα ε, ήθελα να πω ότι η κυρία Ρούλε έχει καλύψει πολλά θέματα και τώρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι διαβολεύσεις μας με τις δημόσιες αρχές στα κράτη δείχνουν ότι συμφωνούν πλέον σε όλους τους διαγωνισμούς να εφαρμόζονται αυτά τα πανενωσιακά κριτήρια. διότι και ο προμηθευτής και ο λεγόμενος έξυπνος πελάτης μπορούν να δεχτούν αυτούς τους κανόνες πια. Έχουν οριμάσει τα πράγματα και γι' αυτό Θέλω και εγώ να συνεργαστώ με τη Χάιντι και να δω τι τροπολογίες θα μπορούσα να καταθέσω και εγώ. Αυτά είχα να πω. Έχουμε λιγάκι καθυστερήσει, αλλά θέλω να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Λόγω όμως των πιέσεων που μα... θα χρειαστεί αμέσως μετά τις διακοπές να ψηφίσουμε. Θέλω να το ξέρετε όλοι λοιπόν, να είστε τηλεγραφικοί και να μην ξαναπείτε πράγματα που έχουν πει και άλλοι. Μάγερ Τσεκόσκι, Στάιλερ, Βάιλερ, Σέρμιν Μέζης και Ρόσφουλ. Κανείς άλλος, Σβάμπ και Γκέμπχαρτ. Παρακαλώ λοιπόν περιοριστείτε στα δύο λεπτά, αλλιώς δεν θα τα καταφέρουμε. Κύριος Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, την κυρία Ρούλε, κυρίως ε, για τις ε, σημερινές ε, προσθήκες ε, τις οποίες θα διαβάσω πολύ προσεκτικά και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κατορθώσουμε να απλουστεύσουμε ουσιαστικά το ευρωπαϊκό δίκαιο ε, ανάθεσης έργων κυρίως να μπορεί να εφαρμοστεί αυτό σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε όλα αυτά που αναφέραμε ε, παραδείγματο χάρη στην οικονομικά ευνοϊκότερη προσφορά αυτό να το ορίσουμε έτσι ώστε να μην παραπέμπονται όλες οι υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο να καλείται να προβαίνει Επίση, Επίσης, ε, θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά ε, και των ε, δημόσιων αρχών. Βεβαίως να υπάρξει βελτίωση αλλά να υπάρχει και μία ασφάλεια τουλάχιστον για τους αναθέτοντες. Επειδή το όλο θέμα αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία όπως και άλλοι συνάδελφοι και εγώ πιστεύω ότι την ηλεκτρονική ανάθεση δεν πρέπει να την προβάλλουμε μόνο στην αιτιολόγηση της έκθεσης. Ε, χάρηκα που άκουσα ότι στην δεύτερη εκδοχή της έκθεσης ε, θα περιλαμβάνεται με ολόκληρη παράγραφος για την ηλεκτρονική ανάθεση. Πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα για τους ε, οργανισμούς εκείνους ε, που θα ασχοληθούν με αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι απλά το να προσφέρονται κίνητρα αυτό δεν είναι αρχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ελπίζω να συζητήσουμε για όλα τα άλλα. Ευχαριστούμε πολύ. Μίλησα για δύο μόνο λεπτά, λέει ο μιλητή. Τσεκόφσκι. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα περιοριστώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν και συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που έκαναν και οι συνάδελφοι. Ιδιαίτερα για την οικονομικά πιο ευνοϊκή προσφορά. Συμφωνώ με τον κύριο Άγκαλ. Για τις μικρές και τις ε, μεσαίες επιχειρήσεις, τα περισσότερα σημεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, που είναι συνοπτική, σε τρεις παραγράφους πιστεύω ότι είναι τα πιο σημαντικά σημεία που μιλάνε για τις, ε, την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό που πιστεύω εγώ ότι λείπει και που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε με μια τροπολογία είναι το θέμα των οικονομικών ε, προϋποθέσεων και συνθήκων όταν υποβάλλουν υποψηφιότητα. Ότι πρέπει να υπάρχει κάποια αναλογικότητα. Γι' αυτό, λοιπόν, χαιρετίζω την έκθεση όσον αφορά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα ήθελα να προσπαθήσω να προσθέσω με κάποια τροπολογία αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε, κυρία Στήλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Θέλω να προσθέσω και εγώ ότι είναι πολύ σημαντικό που μιλάει για την απλοποίηση, για την σαφήνεια η Χάιντι Ρούλε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει όντω να έχουμε βιώσιμε δημόσιε συμβάσει. Αναφέρθηκε στι υπηρεσίε ε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα τις διαφορετικές συνοτροπίες, τις διαφορετικές συνήθειες που υπάρχουν ε, στις διάφορες χώρες. Θέλω να έρθω στο σημείο 19 που αναφέρεται στον επαγγελματισμό. Είναι κάτι που μιλώντας με τους ανθρώπους που δουλεύουν ε, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και που έχουν την πραγματογνωμοσύνη είναι σίγουρα πολύ επαγγελματική και πρέπει να δούμε τι ανταλλαγές μπορούν να υπάρξουν μεταξύ επαγγελματιών του κλάδου ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Θα ήταν ενδιαφέρον να υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με όλους όσοι επένδυσαν την κυρία Ρούλε. Η έκθεσή της είναι σαφής, ε, κατανοητή. Αυτή η δεύτερη εκδοχή διόρθωσε πάρα πολλά. Συμφωνώ και με την πολιτική της ε, τοποθέτηση. Κατά τη διάρκεια των ακροάσεων κατέστη σαφές ότι ήθιστε το δίκαιο συμβάσεων να το χρησιμοποιούν οι ενδιαφερόμενοι σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πολιτικούς και εθνικούς σκοπούς. Και βρίσκω ιδιαίτερα ευχάριστο το γεγονός ότι κατά την ακρόση ε, ο Σύλλογος ε, Βιομηχάνων είπε ότι ως κοινωνικό κριτήριο θα πρέπει να αναφέρεται και η τήρηση των συλλογικών συμβάσεων. Κατόπιν τούτου βλέπουμε ότι έχουμε και συμμάχους ε, που ε, δεν είναι πάντα εύκολο να τους βρούμε. Ε, το βρίσκω πολύ καλό κυρία Ρούλε που ζητάτε απλούς ευέλικτους κανονισμούς και η πρότασή σας ότι η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει σε αυστηρότερο έλεγχο και να προσφέρει και κίνητρα. Σωστό αυτό που λέτε, αλλά δεν θα πρέπει να αγνοούμε τα κράτη-μέλη γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει κάποια αποκέντρωση, τα κράτη-μέλη να μεριμνούν για ταχύ εφαρμογή. Κύριε Μάια, ξέρετε ότι η Γερμανία μόλις πέρυσι εφάρμοσε την οδηγία του 2004 και αυτό αποτελεί σκάνδαλο βλέποντας πόσο σημαντική είναι η οδηγία αυτή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να πω κάτι και για την τιμή κατόφλη. Χαίρομαι πάρα πολύ που η συζήτηση τα τελευταία έξι χρόνια άλλαξε πάρα πολύ. Ε, τώρα γίνεται για την αύξηση σε αυτής τη τιμής, κάτι που εμείς προτείναμε ήδη το 2004. Εν τω μεταξύ όμω, τα πράγματα έχουν αλλάξει στον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για άλλε αγορέ ε, σε ε, παγκόσμιο επίπεδο, παραδείγματο χάρη για την αγορά τη Ινδία. Υπάρχουν ε, συμφωνίε ελεύθερων ανταλλαγών που πρέπει να τροποποιηθούν όπως άκουσα από τους ε, συναδέλφους μου στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου θέλουν ε, οι συνάδελφοι να το ελέγξουν το θέμα, να δουν ε, μήπως το, αν αυξήσουμε τώρα τις τιμές κατόφλι μετά από έξι χρόνια, μήπως αυτό δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΟΕ. Εγώ συμφωνώ, αλλά όχι τελικά ε, να έχουμε προβλήματα. Κυρία Ρούλε, θέλω να γνωρίζω το εξή. Το σημείο 17. Τι ακριβώς εννοείται εκεί. Μήπως εδώ πρόκειται θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα επικίνδυνο κενό και σημείο 21. Αυτό το τροποποίησατε ήδη. Ε, στην πρώτη διατύπωση χρησιμοποίησατε, χρησιμοποίησατε το επίθετο ε, δεσμευτικό. Τώρα όμως το αλλάξατε. Ε, α, ήταν λάθος η μετάφραση. Εντάξει, στα αγγλικά πράγματι ήταν σωστή η διατύπωση, μόνο που η πρώτη γερμανική μετάφραση ήταν λάθος. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα ελέγξετε τις μεταφράσεις τόσο προσεκτικά, γιατί οι μεταφράσεις γραπτές, όταν είναι λάθος, μπορούν να προκαλέσουν πολλά δεινά. Ναι, η κυρία Ρούλε είπε ότι υπάρχει νέα γερμανική εκδοχή. Σαν δε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι και εγώ σύντομη. Δεν θέλω να επανέλθω σε πράγματα που έχουν ήδη υποθεί. Θέλω όμως να προσθέσω το εξής. Όταν συνομίλησα με δανέζικες αρχές και οργανισμούς, ζήτησαν μια αποσαφήνιση των δυνατοτήτων στον κοινωνικό τομέα. Δηλαδή, τι αιτήματα θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε, αναρωτήθηκαν. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό για τη βιωσιμότητα, το πρασίνισμα της οικονομίας. Και μπορεί να πρέπει να υποχρεωτικά να απασχολούμε και εθνικές μειονότητες, ποσοστώσεις δηλαδή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Μπορώ να συνεχίσω από αυτόν που είπε ο Κρίστολ. Γιατί το συζητήσαμε και στην Επιτροπή Απασχόλησης. Δηλαδή, τις δυνατότητες συμπερίληψης της μετεκπαίδευσης για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν. Και να διασφαλίσουμε φυσικά όταν υπάρχουν δημόσιες προμήθειες να εφαρμόζονται και οι συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν. Τρίτον, η συμπερίληψη στοχευμένων ομάδων, προφανές αυτό, και τέταρτον, να διατηρηθούν οι ταξινομήσεις σε α και β για να ικανοποιηθούν και τα κοινωνικά. Να συνδυαστεί δηλαδή η οικονομία με το κοινωνικό θέμα που μερικές φορές το ξεχνάμε και δεν θα έπρεπε. Δεν πρέπει να αντιθέτουμε πάντοτε τα κοινωνικά με τα οικονομικά. Ευχαριστούμε πολύ. Θα φροντίσουμε, θα φροντίσουμε αν και είναι μια απλή γνωμοδότηση. Ο κύριο Ρόσφο. Ροσφόρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ την κυρία Ρούλα για την εκθεσή τη και για να είμαι συγκεκριμένο και σύντομο. θα κάνω δύο σχόλια. Πρώτον, όλοι τελικά συμφωνούμε ότι πρέπει να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και κόστους αλλά πρέπει αυτά να τα βάλουμε σε αριθμούς γιατί να τα πούμε και επίσημα αλλιώς παραμένουν υποκειμενικά θα ήθελα λοιπόν να ζητήσουμε από όλες τις επιτροπές να κάνουν προτάσεις ως προς το τι εννοούν ποιότητα παραδείγματο χάρη αυτά που είπε ο κύριος Κρόιτσμαν προηγουμένως η δυνατότητα δηλαδή όταν ε, γίνεται δεκτή μια προσφορά να βλέπουμε και πώς εφαρμόζεται. Δεύτερον, η διάρκεια όχι της ε, κατασκευής προϊόντων αλλά η διάρκεια των υπηρεσιών που χορηγούνται. Τι εγγυήσεις υπάρχουν πενταετής, δεκαετής. Δεύτερον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αυτές θα ήθελα να προσθέσω ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη δυνατότητα να οργανωθούν μεταξύ τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν οργανώνεται ένας διαγωνισμός μια προσφορά. Δεν πρέπει να, εμποδ... να θεωρηθεί ότι κάτι τέτοιο εμποδίζει ή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Πρέπει να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να οργανώνονται για να έχουν καλύτερες δυνατότητες ανταπόκρισης στο προτινόμενο επίπεδο προσφοράς. Σεβόμενοι βέβαια πάντοτε τον ανταγωνισμό, δηλαδή δεν θέλουμε να καταλήγουμε στη δημιουργία μονοπωλίων, αλλά αν δεν πρόκειται για μονοπόλιο, τότε πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να οργανώνονται. Καλώς οι συντονιστέ μας. Η κυρία Γκέπαρτ πρώτα και μετά ο κύριο Βάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω για αυτό το πολύ καλό σχέδιο το οποίο μας κατέθεσε η κυρία Ρούλη. Μπορούμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά με το σχέδιο αυτό ε, και αυτό είναι ε, κάτι το ιδιαίτερο, όχι ιδιαίτερο όσο την αφορά, αλλά όσον αφορά το αντικείμενο. Κάπως τα μπέρδεψε λέει ο μιλήτρια. Τέλο πάντων ε, ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό το σχέδιο της έκθεσης. Υπάρχει ένα θέμα ε, το οποίο μας απασχόλησε στην αρχή αυτού του αιώνα το θέμα της ε, ευνοϊκότερης ή της ευθυνότερης προσφοράς. Ε, είχαμε πει ότι θέλουμε τη φτηνότερη προσφορά, όμως τα κριτήρια που είχαμε θεσπίσει ήταν λίγο ασαφή. Κατόπιν τούτου προέκυψε νομική ασάφεια, η οποία οδήγησε στο ότι ορισμένα κράτη-μέλη, ορισμένοι αναθέτοντες ε, παρετήθηκαν από τη συμπερίληψη αυτών των ε, κριτηρίων γιατί δεν γνώριζαν κατά πόσον κάτι τέτοιο ήταν νομότυπο ή όχι. Ε, είναι σημαντικό να το διευκρινίσουμε αυτό και αναφέρθηκαν ήδη κάποια παραδείγματα, δεν θέλω να τα επαναλάβω για λόγους χρονικού περιορισμού. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο το βρίσκω εξίσου σημαντικό και το οποίο νομίζω ότι πρέπει να προβάλλουμε περισσότερο είναι ότι δεν πρέπει να αφήσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να νομοθετήσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τους πολιτικούς τομείς. Εδώ αναφέρομαι κυρίως στις συμβάσεις παραχώρησης. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ε, καθίστανται απαραίτητες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γιατί πολλοί δεν γνωρίζουν ε, τι ακριβώς είναι αυτές οι συμβάσεις παραχώρησης. Αυτό όμως είναι σημαντικό. Ξέρω ότι εδώ διαφωνούμε λιγάκι με την κυρία Ρούλε επί του πράγματι θα πρέπει το θέμα αυτό να το συζητήσουμε περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σουάπ. Ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Ε, πιστεύω ότι η έκθεση της ε, κυρίας Ρούλε θέτει τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Δηλαδή προσπαθεί να εξετάσει τα θέματα εκείνα που ενδείκνυνται για κάποια αλλαγή. Κατόπιν τούτου η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Το ΕΛΚ ε, θα στηρίξει ε, πολλά σημεία της έκθεσης, όπως ήδη είπε η κυρία Έγγελ. Εγώ προσωπικά στηρίζω ιδιαίτερα αυτό τον ε, συνετό τρόπο εξέτασης της αλλαγής της τιμής κατόφλη. Διότι, όπως είπε η κυρία Έγγελ, δεν πρέπει να περιζόμαστε μόνο στις ε, δικές μας ε, τις ε, αγορές, αλλά θα πρέπει να έχουμε κατά νου και τις εξαγωγές στον υπόλοιπο κόσμο. Δεύτερον, στηρίζω ιδιαίτερα αυτή την έννοια της ευνοϊκότερης προσφοράς. Πολύ σωστά όσα ελέγχθησαν από αυτού. Βέβαια πρέπει να το διευκρινίσουμε λιγάκι, γιατί δεν αρκεί απλά το να το συζητάμε θεωρητικά. Εκεί που διαφωνούμε λιγάκι είναι αφενός Μάλλον, συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα τη απλούστευση των διαδικασιών, μόνο που τίθεται το ερώτημα κατά πόσο αυτό είναι εύκολο να γίνει. Ε, θέλω να σα υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόσφατα ε, στην απόφαση Arnhorn ε, κατέθεσε και ξεκαθάρισε περισσότερο ένα σημείο που για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ασαφέ. Όταν όμω αλλάζουμε συνεχώ ε, την ομολογία, τελικά δεν επιτυγχάνουμε απαραίτητα νομική σαφήνεια, αλλά δημιουργούμε κάποια σύγχυση. Τελευταία μου παρατήρηση. Και εδώ πρέπει να πω, συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φρανκ Έγγελ, ε, δηλαδή η εισαγωγή της ε, στάνταρ διαδικασίας δεν είναι πάντα ο καλύτερος δρόμος. Και εδώ ε, πρέπει να υπάρξει κάποια απλούστευση και μένει ανοιχτό το να δούμε πώς θα το επιτύχουμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την τόσο καλή συζήτηση. Κύριε Σμιτ, τώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο. Θέλετε να απαντήσετε σε κάποια σημεία σύντομα και μετά θα δώσω το λόγο στην κυρία Ρούλε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ, κύριε Σμιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως πάντα, θα σας πω και τώρα ότι τα άκουσα όλα, τα σημείωσα. Χαιρόμαστε που διαπιστώνουμε ότι συμφωνούμε σε πάρα πολλά σημεία και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε κάτι που θα ικανοποιεί την ΙΜΚΟ, την Επιτροπή σας. Θέλω όμως να υπογραμμίσω το εξή. Μία προειδοποίηση για το κατόφλι αλλά και για την απλοποίηση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε διεθνείς υποχρεώσεις. Όσον αφορά τις ε, δημόσιες συμβάσεις δεν πρόκειται μόνο για το κατόφλι, πρόκειται και για διαδικασίες οι οποίες έχουν συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε όταν προχωρήσουμε και καταλήξουμε στις διαδικασίες. Εννοείται ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στα πλαίσια αυτών των συμφωνιών. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ για την συμβουλή που μας δίνετε. Θα την έχουμε υπόψη μας. Τώρα η Χαϊντή Ρούλε για να ολοκληρώσει και να μας επιβεβαιώσει και το χρόνο διάγραμμα, έτσι. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι ε, σκιώδεις ε, συντονιστές δέχτηκαν ότι τώρα πρέπει να τεθεί ε, η προθεσμία ε, γιατί αν αυτό μετατίθετο, δηλαδή αν μετατίθετο η 19 η Ιουλίου θα υπήρχε πρόβλημα. Γι' αυτό και εγώ προσπάθησα να διορθώσω στο συντομότερο δυνατόν τη γερμανική μετάφραση για να μπορείτε να τη δουλέψετε. Ε, όλοι οι συνεργάτες έχουν τις δικές μου τις ε, τροπολογίες αλλά θα σας τις στείλω τις ε, τροπολογίες αυτές στα αγγλικά και σε όλους σας να τις έχετε, να τις γνωρίζετε έτσι ώστε πάνω σε αυτές να μπορείτε και εσείς να στείλετε τις δικές σας τροπολογίες. Και όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Βάλερ θα τα κουβεντιάσουμε σε διμερές επίπεδο. Κατά τα άλλα ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συζήτηση και χαίρομαι και προσβλέπω στις τροπολογίες σας. Ευχαριστούμε πολύ. Προθεσμία είναι η 19η Ιουλίου για την κατάθεση τροπολογιών. 19 Σεπτεμβρίου θα συζητήσουμε και θα ψηφίσουμε στην ΕΜΚΟ. Και στην δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου, λέει ο Πρόεδρος, θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια την τελική πρόταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συνεχίζουμε και περνάμε στην επόμενη έκθεσή μας. Έχουμε σχέδιο έκθεσης εδώ. Της κυρίας Χάντσλικ για τη διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση σύμφωνα με την οδηγία για τι υπηρεσίε. Οι σκιώδε είναι εδώ, κύριε Κέπερτ, ο κύριο Μάντερ. Ο κύριο Κάνφα είναι εδώ. Ή μιλάει κάποιο άλλο εκ μέρου των Πρασίνων. Όχι, εγώ είμαι εδώ. Οι υπόλοιποι δεν είναι εδώ. Και ο Μάρτιν Φρόν εδώ από την Επιτροπή. Ναι. Ωραία. Θα δώσω το λόγο λοιπόν στην κυρία Χάντσλεκ πρώτα απ' όλα για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της και μετά θα ακούσουμε τους υπόλοιπους. Έχουμε καθυστερήσει λίγο, αλλά ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο για συζήτηση. Και η κυρία Σβέντσεν εδώ για την επόμενη έκθεση που έχουμε. Παρακαλώ κύριε Χάντσλικ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η οδηγία για τις υπηρεσίες είναι μία πολύ βασική νομοθετική πράξη, από τις πιο βασικές που έχουμε συζητήσει εδώ στην Επιτροπή αυτή. Και εξακολουθούμε να τα βάζουμε με την οδηγία αυτή και πρόσφατα μάλιστα και επί τη ευκαιρία της έκθεσης αυτής. Τώρα όμως και στα πλαίσια της διαδικασίας αμοιβαία αξιολόγησης. Είναι μια διαδικασία η οποία προβλέπεται από το άρθρο 39 Τη οδηγία. Πρόκειται για ένα νέο μέσο που έχουμε στη διάθεσή μα και που χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διαδικασία μηδέα αξιολόγησης δεν καλύπτει, πρέπει να ξέρετε, όλα τα άρθρα της οδηγίας, αλλά ασχολείται με ορισμένες μόνο προϋποθέσεις, ορισμένες διατάξεις, οι οποίες επιτρέπουν ε, στα κράτη-μέλη να έχουν ένα βαθμό διακριτικής ευχέρειας. Η δομή της έκθεσής μου απορρέει από τις συζητήσεις που έγιναν στα εργαστήρια για τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης και καλύπτει ιδιαίτερα τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα, την εμπειρία που έχουμε συσσωρεύσει όσον αφορά τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης για την οδηγία για τις υπηρεσίες τα αποτελέσματα και τις δράσεις βάσει αυτών. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι η αμοιβαία αξιολόγηση ως μέσο για τις μελλοντικές νομικές πράξεις. Στην έκθεσή μου υπογραμμίζω ότι η αμοιβαία αξιολόγηση δεν ε, πρέπει να είναι κάτι που την μπερδεύουμε με την διαδικασία εφαρμογής. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγησης δεν έχει ως στόχο την βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας, αλλά την αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά την ενιαία αγορά, τις υπηρεσίες δηλαδή στα πλαίσια της ενιαίας αγοράς. Η διαδικασία αυτή αμοιβαίας αξιολόγησης έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε, εφαρμογής. Μια προπόθεση η οποία δεν έχει καλυφθεί όμω πλήρω όσον αφορά την οδηγία για τι υπηρεσίε. Οι καθυστερήσει που υπάρχουν στην εφαρμογή τη οδηγία μπορεί να έχουν επηρεάσει και την διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση. Πάντω πιστεύω ότι η διαδικασία αμοιβαία αξιολόγηση είναι κάτι που πρέπει να το βλέπουμε σαν ένα στοιχείο κλειδί ενίσχυσης της Διαδικασία διοικητική συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών και ε, βοηθάει στην ε, καλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των υπηρεσιών. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο αξιολόγησης που μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τα μελλοντικά εμπόδια της ενιαίας αγοράς στον τομέα των υπηρεσιών. Η διαδικασία αυτή είναι μία προστιθέμενη αξία το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα του τι γίνεται στα κράτη-μέλη όσον αφορά τις προϋποθέσεις που εμπίπτουν στη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης. Και χτυπάει το κουδουνάκι όσον αφορά τη διαφάνεια. Τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης, αλλά είναι πράγματα τα οποία ακούγονται στη δημόσια διαβούλευση που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε αυτή τη διαδικασία πάντως αυτό το οποίο ε, λείπει είναι οι τακτικές εκθέσεις. Μετά από κάθε συνάντηση δηλαδή τι συμπεράσματα έχουμε. Συμπεράσματα στα οποία να μπορούν τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση. Αυτή η πτυχή της διαδικασίας θα μπορούσε να βελτιωθεί στο μέλλον όσο δηλαδή περισσότερο χρησιμοποιούμε τη διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης. Αυτή η διαδικασία έχει χρησιμοποιηθεί και για άλλες πράξεις που χρησιμοποιεί στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αξιολογήσει γενικότερα την αγορά εσωτερικών, την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για τις συζητήσεις που γίνονται με τα κράτη-μέλη. Έχω την εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να ενημερώνεται για τις συνομιλίες αυτές. Έχω όμως την αίσθηση ότι χάνουμε τη γενικότερη εικόνα και οι περισσότεροι από εμά πολύ θα θέλαμε να έχουμε πληροφορίες όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής. Έπειτα, ο χρόνος που πέρασε από την εφαρμογή της οδηγίας επηρεάζει κατά πολύ τις προϋποθέσεις πλήρους εφαρμογής της οδηγίας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή φαίνεται να προτείνει και μια διαδικασία ε, αξιολόγησης επιδόσεων Οι δράσεις που προωθούν τις υπηρεσίες της ενιαίας αγοράς πρέπει να επικεντρώνονται στους τομείς εκείνους όπου υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατότητα διασυνοριακών ανταλλαγών. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τις διατάξεις της διαδικασίας αμοιβές αξιολόγησης. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει διάφορα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις υπηρεσίες όσον αφορά ε, τις κεφαλαϊκές αγορές, για παράδειγμα, ή τα θέματα ασφάλειας. Γι' αυτό και προτείνω αυτά τα θέματα να τα κοιτάξουμε περισσότερο είναι προβλήματα τα οποία έχει εντοπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο στα πλαίσια της οδηγίας για τις υπηρεσίες αλλά και αλλού και ζητάει δράση από τη δικιά μας την πλευρά. Η έκθεσή μου επίσης θίγει και ένα άλλο θέμα. Την οικονομική εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, κάτι το οποίο έχει ήδη αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σύνολο της διαδικασίας αμοιβές αξιολόγησης. Πάντως πιστεύω ότι πρέπει να τύχει της υποστήριξής μας. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται για τα όσα συμβαίνουν. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες μας από τη διαδικασία αμοιβέ αξιολόγηση και σε άλλους πολιτικούς τομείς. Συστήνω λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό αξιολόγησης και στο μέλλον βέβαια υπό προϋποθέσεις. Πιστεύω ότι η αμοιβαία αξιολόγηση πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως σε οριζόντια μέτρα, τα οποία να προστατεύουν τα κράτη-μέλη. Τέλος, η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για στοιχεία κλειδί ε, των οδηγιών και όχι γενικότερα. Να χρησιμοποιείται δηλαδή πιο συχνά, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς που τους έχουμε αναλύσει προηγουμένως πολύ και τα διαφερόμενα μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται για την πρόοδο των εργασιών. Εν κατακλείδη, πιστεύω ότι η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης αποτελεί ένα καλό μέσο, παρόλο που έχει και τις αδυναμίες του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε νέους τομείς. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε δράσεις που βελτιώνουν την εσωτερική αγορά υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει την πρόταση ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς. Όμως, ο πρώτος και κύριος στόχος μας παραμένει η ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο προς το παρόν περιμένω να ακούσω τα δικά σας σχόλια. Ιδιαίτερα από τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χάνσλικ. Τώρα θα ακούσουμε τους σκιώδεις, η κυρία Γκέμπχαρτ πρώτη. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Χάνσλικ ε, για το πολύ ωραίο σχέδιο έκθεσης που καταθέσατε όπου εξετάζεται ένα θέμα ε, για το οποίο συζητήσαμε διαμακρών όταν ασχοληθήκαμε με την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Τότε λοιπόν ε, στο Κοινοβούλιο η συντριπτική πλειοψηφία έκρινε ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό μέσο το οποίο το απορρίψαμε όμως τα κράτη-μέλη είπαν εμείς το επιθυμούμε και εμείς ε, ανταπαντήσαμε ότι εντάξει θα δούμε τι θα γίνει και πώς ακριβώς λειτουργεί. Νομίζω οι αρχικές επιφυλάξεις που είχαμε ως ε, Κοινοβούλιο, οι επιφυλάξεις αυτές ε, φάνηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δικαιολογημένες. Καλό αυτό γιατί μαθαίνουμε πράγματα και νομίζω ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν σωστή. Δηλαδή παρουσιάστηκαν μικρές ομάδες ε, κρατών και δεν έπρεπαν όλοι να ενημερωθούν για όλα. Επιλέχθηκε λοιπόν μια διαδικασία που είναι λογική και που οδηγεί στο στόχο. Οδηγεί στο στόχο κυρίως ε, με την εξή έννοια. Έχω την εντύπωση ότι η διαδικασία αυτή συνέβαλε στο ότι ορισμένοι φόβοι που υπήρχαν στη διοίκηση για πολίτες από άλλες χώρες και με άλλους ε, πολιτισμούς ε, η άγνοια που υπάρχει σε ορισμένα κράτη ξεπερνιέται πολύ πιο εύκολα και με τον τρόπο αυτό παρισφρεί στη διοίκηση περισσότερο το ευρωπαϊκό στοιχείο. Αν αυτό είναι ένας από τους στόχους ε, που θέλαμε να πετύχουμε και αν τον πετύχαμε, πετύχαμε πράγματι πάρα πολλά. Κατόπιν τούτου ο τρόπος προσέγγισης είναι σωστός. Βεβαίως έχετε δίκιο ε, λέγοντας ότι αυτό δεν μπορεί να το εφαρμόζει παντού γιατί πράγματι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό εργαλείο. Κατόπιν τούτου στο μέλλον ε, αν ε, εφαρμοστεί το εργαλείο αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε να δούμε πού και πώς θα εφαρμόζεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θα ήθελα να το δω να προβάλλετε περισσότερο στην έκθεσή σας. Δηλαδή να εφαρμόζεται το εργαλείο αυτό ε, σε πραγματικά περίπλοκα ζητήματα και όχι γενικότερα ε, στην γενικότερη νομοθεσία. Ε, γιατί εγώ στη γενικότερη νομοθεσία το που κρίνω σωστό είναι να υπάρχουν πίνακες αντιστοίχησης για να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς ακριβώς εφαρμόζονται οι νόμοι. Και αυτό το σημείο θα ήθελα να το προβάλλετε περισσότερο στην έκθεσή σας. Ναι, μεν το αναφέρετε, αλλά θα επιθυμούσα, όπως σας είπα, να προβάλλετε περισσότερο το στοιχείο αυτό. Πέρα από όλα αυτά τα ιδιαίτερα θετικά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να σκεφτείτε ε, το κατά πόσον ε, τα σημεία 16 και όσα ακολουθούν ε, θέλετε να τα αφήσετε στην έκθεση σας ή όχι γιατί αυτά αφορούν ε, την αξιολόγηση της οδηγίας παροχής υπηρεσιών και όχι την, ε, τη διαδικασία αξιολόγησης, αμοιβαίας αξιολόγησης αυτό το έκανα και εγώ στη δική μου την έκθεση, δηλαδή να μην ξεκινήσουμε συζήτηση επί της ουσίας. Ε, νομίζω ότι ίσως μπορείτε να το σκεφτείτε λιγάκι αυτό, ε, το άρθρο 16 και όσα μετά ακολουθούν, κατά πόσον θέλετε να τα διατηρήσετε ή όχι. Γιατί αν τα διατηρήσετε, η συζήτηση ε, θα δυσχέρανθει. Το θέμα αυτό κατά κάποιον τρόπο ξεπερνάει το αντικείμενο της εκθεσίας και πρέπει λιγάκι να το συζητήσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε με τα θέματα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Μάθιος. Ευχαριστώ. Η οδηγία των υπηρεσιών θα έπρεπε να είναι από τους ακρογωνιαίους λίθους γενικά των προγραμμάτων μας. Ευτυχώς λειτουργεί μέχρι τώρα σωστά. Εγώ είμαι υπέρ των ιδεών που εκφράζονται εδώ, αλλά φοβάμαι ότι στην πράξη δεν θα εφαρμοστούν σωστά. Όπως είπα πρέπει να είναι ακρογωνίος λίθος καθώς και η ελεύθερη διακίνηση, αλλά τα κράτη-μέλη προσπαθούν να προστατεύσουν το καθένα τις δικές του υπηρεσίες και προμηθευτές. Και αν το κάνουν αυτό όλα τα κράτη θα ξαναδημιουργήσουμε σύνορα εσωτερικά. Κρίμα. Είμαι όμως υπέρ της ιδέας δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που είπαν άλλοι ομιλητέ και η δήλωση της Κομισιόν είναι κατ' εμέ πολύ αισιόδοξη. Κι εγώ όμως είμαι αισιόδοξο. Αν εφαρμοστούν σωστά όλα αυτά θα ήμουν πολύ ικανοποιημένο, αλλά βλέπω ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία μέχρι τώρα και αυτό κρίμα. σχεδόν τίποτα δεν άλλαξαν στην νομοθεσία τους για να καταργήσουν απαράδεκτους φραγμούς και γι' αυτό βλέπετε ότι προστατευτικά μέτρα, προστατευτιστικά μέτρα υπάρχουν ακόμη. Όταν η Εύελιν και εγώ δίναμε τη μάχη για το θέμα αυτό, εξαιρέσαμε ορισμένους τομείς και μέχρι τώρα δεν έχουν τύχει εναρμόνισης όπως οι υγειονομικές υπηρεσίες κλπ. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συμπεριληφθούν κάποτε και αυτοί. Στη νομική επιτροπή έγινε ψηφοφορία και πάλι επιδείχτηκε εκεί εθνικιστικό πνεύμα. Είναι δύσκολο να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Χαίρομαι όμως ιδιαίτερα γιατί υπάρχει αυτή η ιδέα της single contact. Δεν ξέρω τι προστίθεται τώρα εφόσον υπάρχουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ήδη. Αν και είναι μάλλον βέβαιο ότι δεν συμπεριφέρονται όλα τα κράτη όπως θα έπρεπε. Και αυτό αν εφαρμοστεί θα ήμουν πολύ ικανοποιημένος ίσως σε 5, 6, 10 χρόνια όταν θα είμαστε πια στη σύνταξη να πούμε ότι δουλεύει επιτέλους σωστά. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ε, χαρακτηριστικά πολεμική σας ε, τοποθέτηση. Τώρα θα μιλήσω εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου. Α, ήθελες Χάιντι να προσθέσεις τίποτα. Πολύ σύντομα θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση στον ε, προλαλήσαντα. Κύριε Μάντες, ε, ίσως ε, θα έπρεπε να διαβάσετε την έκθεση του συναντέλφου σας από την πολιτική ομάδα σχετικά με τα ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια που αυτός έχει άλλη άποψη από εσάς. Τέλος πάντων, εγώ ζήτησα το λόγο για, άλλο λόγο. Αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση θεωρώ ότι είναι μια καλή προσέγγιση. Η κυρία Χάνσλικ παρουσίασε το θέμα πολύ σωστά ε, μόνο που στο επεξηγηματικό σημείωμα ε, κάνει την παρατήρηση ότι πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις σημαντικότερες ε, διατάξεις και το λέει αυτό για να αποφύγει να προκύψει περιττή γραφειοκρατία. Το βρίσκω αυτό πολύ σωστό στην ε, αιτιολογική της έκθεση ε, και θα ήταν καλό να περιλαμβάνεται και στο κύριο σώμα της οδηγίας. Ε, αυτό έχει πάλι να κάνει με την εφαρμογή στα κράτη-μέλη, γιατί πήραμε πάρα πολλές προσφυγές από την τοπική αυτοδιοίκηση στη Γερμανία και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την εφαρμογή. Το πώς εφάρμοσε η γερμανική κυβέρνηση αυτή την οδηγία. Κατά τα άλλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκθεσή σας. Και εγώ αυτά ήθελα να πω. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ να ξανασυζητήσουμε το θέμα του εύρους της οδηγίας των υπηρεσιών. Νομίζω όμω, όπως είπε και η κυρία Χάνσρικ, ότι η σημασία εδώ έγκυται στην εφαρμογή μιας πολύπλοκης νομοθεσίας για την ενιαία αγορά έγκυται στην εφαρμο... <laughs> στη δυσκολία εφαρμογής μιας πολύπλοκης νομοθεσίας για την ενιαία αγορά. Το όλο θέμα της οδηγίας των υπηρεσιών ήταν ότι τα κριτήρια για τις απαλλαγές ορισμένων τομέων είχαν συζητηθεί πάρα πολύ. Βλέπω ότι χαμογελάει η κυρία Γκέπχαρτ γιατί το ξέρει το θέμα οι διαπραγματεύσεις για το άρθρο 16 ήταν μακροσκελέστατες και το θέμα σήμερα για την ενιαία αγορά είναι πώς θα υπάρξει κάποια συνοχή μεταξύ και συνδυασμός μεταξύ αυτών που θέλουν οι εθνικές αρχές και το άρθρο 16. Η πρόοδος που έχει συμβεί εδώ για την αξιολόγηση της εφαρμογής της οδηγίας είναι ότι και τα ίδια τα κράτη-μέλη μεταξύ τους χρειάστηκε να συνεννοηθούν. Είχαμε πει ότι πρέπει να γίνεται περισσότερη αμοιβαία αξιολόγηση όπως για τις τηλεπικοινωνίες αντί με κεντρικό τρόπο από την Κομισιόν. Αλλά σε αυτό επέμεινε πολύ το κοινόβουλιο και το ότι γίνεται πια αυτή η αμοιβαία αξιολόγηση νομίζω είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά συμφωνώ και πάλι με αυτά που είπε η κυρία Χάνσλικ ότι δεν πρόκειται για εργαλείο πανάκια για κάθε περίπτωση. Χρειάζεται εδώ κάποια κρίση και τα θέματα της αμοιβαία αξιολόγηση ορισμένων αγαθών είναι αντικείμενο περιορισμών ακόμη από ορισμένα κράτη-μέλη και για τη διαμεθοριακή τους διακίνηση. Γιατί μερικά κράτη-μέλη θεωρούν προϊόντα επικίνδυνα που άλλα κράτη-μέλη δεν τα θεωρούν επικίνδυνα. Χρειάζεται λοιπόν μεν περισσότερη αμοιβαία αξιολόγηση αλλά και περισσότερος διάλογος μεταξύ των χωρών μελών. Γιατί Μπορεί μια χώρα να απαγορεύει μια υπηρεσία ή ένα αγαθό για λόγους ε, συμφέροντος των πολιτών της, ενώ η ίδια υπηρεσία ή αγαθό πωλείται ή χορηγείται ελεύθερα στη διπλανή χώρα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί. Τέλος για αυτά που είπε η κυρία Γκέπχαρτ συμφωνώ ότι δεν είναι η καταλληλότερη στιγμή και χώρος εδώ για να λύσουμε εδώ τα προβλήματα στην εφαρμογή της οδηγίας των υπηρεσιών αλλά έχει δίκιο ότι τα συμπεράσματα των αμοιβαίων αξιολογήσεων είναι πολύ ενδιαφέροντα γιατί δείχνουν πόσο πολύπλοκα είναι τα θέματα αυτά. Για μένα ήταν απρόσμενο, απροσδόκητο ότι οι υποχρεώσεις ασφάλισης εφαρμόζονται για ορισμένους χορηγούς υπηρεσιών μεταξύ χωρών μελών ενώ η ασφάλιση υπάρχει ήδη από τη χώρα προέλευσης. Αυτό μου φαίνεται προβληματικό γιατί πρόκειται για έλλειψη εμπιστοσύνης. Κάποιος που είναι ασφαλισμένος σε μία χώρα θεωρείται δηλαδή ότι δεν είναι ασφαλισμένος στην άλλη γιατί δεν έχουν, γίνει απαραί... δεν έχουν ανταλλαγή, ανταλλαχθεί οι απαραίτητες πληροφορίες για να λειτουργήσει καλά η ενιαία αγορά. Και επίσης η... να δίνονται μόνο σε ορισμένους επαγγελματίες, ορισμένες υπηρεσίες είναι και αυτό προβληματικό. Καλό είναι που το ταυτίσαμε και πρέπει να ζητήσουμε για αυτά τα θέματα να μας τα εξηγήσει η Κομισιόν. Τώρα τι λύσεις θα μας προτείνει είναι πολιτικό πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον να τα ταυτίσουμε και να τα θέσουμε. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εγώ για την έκθεσή σας. Και ερχόμαστε τώρα με καθυστέρηση στο θέμα του Μάρτιν Φέλμς. αν έχει να μας κάνει κανένα άλλο σχόλιο πριν λήξει αυτό το θέμα για κάνα δυο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομα γιατί ξέρω ότι υπάρχει καθυστέρηση. Μερικά σχόλια λοιπόν Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ικανοποιημένοι από την έκθεση αυτή. Νομίζουμε ότι θέτει τα σωστά θέματα και με βάση την εμπειρία μας από το άρθρο 39 της Οδηγίας των Υπηρεσιών τα αποτελέσματα, τα κριτήρια δεν ήταν και πολύ ενθαρρυντικά. Προσπαθούμε λοιπόν να τα ενισχύσουμε και με χαρά άκουσα ότι η κυρία Γκέμπχαρτ αναγνωρίζει ότι είναι ωφέλιμη, χρήσιμη αυτή η διαδικασία αξιολόγησης και όχι άχρηστη γραφειοκρατία. Συμφωνούμε όλοι ότι, λοιπόν ότι είναι χρήσιμη η αξιολόγηση. Επίσης, καλό θα ήταν όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε να τονιστούν και τα συμπεράσματα από την ανακοίνωσή μας γιατί νομίζουμε ότι έτσι φαίνεται πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμη περαιτέρω η λειτουργία της οδηγίας των υπηρεσιών. Συμφωνώ απόλυτα και για όσα υπόθηκαν για την περιορισμένη χρήση που πρέπει να γίνεται ορισμένων εργαλείων αμοιβαίας αξιολόγησης μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα αλλά πρέπει και να χρησιμοποιείται σωστά. Δεν είναι καθημερινό εργαλείο. Είναι για έκτακτες και σοβαρές περιπτώσεις. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε κοινό στόχο με το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάνσλικ για να συμπεράνει. Η διορία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 18 Ιουλίου και μετά τις διακοπές στις 31 Αυγούστου ελπίζω να είστε όλοι παρόντες και όλες παρούσες για να δούμε τις τροπολογίες και μετά να τις ψηφίσουμε στις 19 Σεπτεμβρίου και με κατάσταση στην Ολομέλεια. Η ε, κύριε Χάντκιν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά σας. Γενικά βλέπω ότι συμφωνούμε για το ότι η διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης αποτελεί ένα καλό μέσο, αλλά ένα μέσο το οποίο δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε παντού και πάντα, πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν και όπου μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για οριζόντιες οδηγίες, μόνο για οριζόντιες ε, οδηγίες. Και από ό,τι βλέπω συμφωνείτε μαζί μου από αυτού. Κατά τα άλλα, ε, σημειώνω και συμφωνώ με τις περισσότερες από τις παρατηρήσεις σας που θα συζητήσω διμερώς με τους συναδέλφους εδώ για να δούμε πώς μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Οι νέες τροπολογίες θα δώσουν μια νέα διάσταση και θα βελτιώσουν αναμφίβολα το περιεχόμενο της έκθεσής μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων για τη συνεργασία σας και σας εύχομαι επί τη ευκαιρία καλές διακοπές. Thank you very much. ευχαριστούμε πολύ. Σίγουρα θα έχετε χρόνο να διαβάσετε τις τροπολογίες μας. Έχετε χρόνο με τις διακοπές. Και τώρα περνάμε στο τελευταίο μας θέμα για σήμερα το απόγευμα και χαίρομαι πολύ που έχουμε εδώ την εισηγήτρια για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων, είναι η κυρία Εύα Μπριτ Σφένσον και πρόκειται για μια νέα στρατηγική για την πολιτική προστασία των καταναλωτών. Θα σας δώσω το λόγο. Έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Λοιπόν, θα έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψε, ξέροντας ότι θα επανέλθουμε στο θέμα έτσι κι αλλιώς. Η κυρία Λεγκρίπ είναι εδώ από τους Σκιώδης. Για τον κύριο Ρέπο ποιος. Α, η κυρία Γκέπαρ θα μιλήσει, ο κύριος Ροσφόρ, η κυρία Ρούλε έφυγε, ελπίζω να γυρίσει. Εγώ πάλι εκ μέρους του ECR και ο κύριος Σαλβίνη. Ωραία, άρα έχουμε full house. Και χαίρομαι πολύ που έχουμε εδώ και την κυρία Ζάκλεν Μάινερ και την κυρία Σκημισού που είναι δύο από τους πιο υψηλούς στην ε, ΣΑΝΚΟ και δικαιοσύνη. Συγγνώμη που δεν τα είπα όλα. Η κυρία Μισού είναι γνωστή σε εμά από τη δουλειά της ανθρώπινα δικαιώματα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε και οι δύο εδώ θα σας ακούσουμε, έστω και σύντομα θα σας ακούσουμε πριν ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Κυρία Σβένσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να δουλέψω μαζί με τους συναδέρφους πάνω στη στρατηγική για την πολιτική προστασία των καταναλωτών. Λοιπόν, είχα σκεφτεί να παρουσιάσω τις προτεραιότητές μου στους συναδέρφους και από εκεί και πέρα να ακούσω τις απόψεις των συναδέρφων και να τις σημειώσω βέβαια. Ξεκινάω λέγοντας ότι αυτή η στρατηγική υπέρ των καταναλωτών είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες, είναι πολύ χρήσιμο για αυτούς. Βλέπετε μεταξύ των καταναλωτών, των συμπολιτών μας, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για τις επιχειρήσεις. Τώρα όμως έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε και στον κάθε Ευρωπαίο πολίτη ότι έχουμε κάτι που είναι προς όφελος των ίδιων των καταναλωτών. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτήν την ε, οπτική γωνία πάντα από την πλευρά των καταναλωτών. Η κυρία Ρέντινγκ, η Επίτροπος Ρέντινγκ, την άνοιξη του 2012 θα παρουσιάσει μια νέα ατζέντα για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Στόχος είναι να καταδείξουμε ότι στην νομοθεσία υπέρ των καταναλωτών συμπεριλαμβάνονται όλα. Εμείς στο Κοινοβούλιο θέλουμε και χαιρόμαστε για αυτήν την υψηλή φιλοδοξία της Επιτρόπου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς του Κοινοβουλίου έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα να περάσουμε και τις δικές μας απόψεις και να συμπεριλάβουμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους καταναλωτές. Καλό λοιπόν θα ήταν να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μεγάλη πλειοψηφία που στηρίζει την στρατηγική αυτή. Όταν ε, εισήχθη η νομοθεσία υπέρ των καταναλωτών, πρόκειται κυρίω για θέματα που είχαν να κάνουν με τη διατροφή, με την υγεία, με την ασφάλεια. Σίγουρα αυτά βρίσκονται πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη, αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μα. Πρέπει να προστατεύσουμε, για παράδειγμα, τα παιδιά από τι διαφημίσει. Υπάρχουν επίσης χημικά που χρησιμοποιούνται και που είναι ευλαβερά για την υγεία. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική λοιπόν για τους καταναλωτές που θα συνεισφέρει επίσης στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής του 2020. Μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα για παράδειγμα. Η αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης, της ψηφιακής οικονομίας ή επίσης γύρανση του πληθυσμού. Πρέπει να μειώσουμε επίση τα χάσματα και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν διαφορετικές καταστάσεις ε, ανάλογα με το σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Στο κάτω-κάτω δεν είμαστε μόνο καταναλωτές, είμαστε και πολίτε, είμαστε άνθρωποι. Δεν πρέπει να μας περιορίζουν μόνο στην ιδιότητα του καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη ισχύ στις οργανώσεις καταναλωτών τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θέλω επίσης να πω ότι έχοντας υπόψη μας το βαθμολόγιο όσον αφορά ε, τους καταναλωτές υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο που δεν έχουν πρόσβαση σε πολύ βασικές πτυχές της ζωής. Και έχουμε συγχρόνως και καταναλωτές οι οποίοι έχουν πάρα πολλές σπόρους στη διάθεσή τους. Δουλειά μας είναι να φέρουμε κάποια ισορροπία στην κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε να χτίσουμε μια κοινωνική Ευρώπη με κοινωνικές υπηρεσίες στις οποίες θα έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Άρα λοιπόν ας δράξουμε την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται. Υπάρχουν βέβαια αρχέ της Λισαβόνας που λένε ότι οι πτυχές του καταναλωτή είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Και πώς επίσης θα έχουμε μια βιώσιμη οικονομία και για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες και πώς θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών όταν για παράδειγμα κάνουν αγορές μέσω του διαδικτύου. Πώς θα είναι ενημερωμένοι οι καταναλωτές έτσι ώστε τα δικαιώματά τους να προστατεύονται πλήρως. Τρεις είναι οι προτεραιότητες πάνω στις οποίες θέλω να βασιστώ. Βιωσιμότητα, ασφάλεια και προστασία των παιδιών μας από τις διαφημίσεις. Βάσει της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, η Ευρώπη θέλει να φτιάξει, να έχει μάλλον στη διάθεσή της μια ανάπτυξη, η οποία να είναι ευφυής και η οποία να βοηθήσει να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι πολίτες αυτήν, να υποφελούνται όλοι οι πολίτες από αυτήν. Η στρατηγική μας λοιπόν πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι η ιδιωτική κατανάλωση θα βοηθήσει την επίτευξη των στόχων αυτών. Οι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα από την παραγωγή ενέργειας ή από τις μεταφορές αυξάνονται συνεχώς στην Ευρώπη και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας στη στρατηγική μας για τους καταναλωτές. Επίσης, 90 εκατομμύρια τόνοι τρόφιμα ε, πετιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να ε, συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Το 2050 εξάλλου η ζήτηση στα τρόφιμα θα αυξηθεί κατά 70% παγκοσμίω. Και εδώ πρέπει να ευθυγραμμιστούμε λοιπόν με ε, με την κατάσταση, με την πραγματικότητα και να το λάβουμε αυτό υπόψη μας στη στρατηγική μας για τη γεωργία. Ασφάλεια τροφίμων τώρα και ασφάλεια προϊόντων είναι και αυτός ένας τομέας όπου οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα χημικά. Επί παραδείγματι, στα διάφορα προϊόντα που καταναλώνουμε καθημερινά. Εδώ χρειάζεται επίσης μεγάλη προστασία των καταναλωτών. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που απασχολούν τους πολίτες μαζί με την ασφάλεια τροφίμων και την ρύθμιση των ε, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η στρατηγική μας για τους καταναλωτές επίσης πρέπει να υποστηρίζει υγιεινές εναλλακτικέ, να έχουμε επίσης πολύ καλή σήμανση στα προϊόντα μας. Αλλά δεν πρόκειται μόνο για το θέμα της σήμανσης, τι αναφέρουν οι ετικέτες πάνω στις συσκευασίες. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και έτοιμοι να απαγορεύσουμε ουσίες οι οποίες ξέρουμε ότι είναι επικίνδυνες για την υγεία μας. Είναι μια ευθύνη πολύ μεγάλη για μας και πρέπει να την παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Κάτι άλλο επίσης είναι ότι το σύστημα Ripex πρέπει να είναι πιο διάφανο και πιο αποτελεσματικό, έτσι ώστε οι καταναλωτές να ξέρουν ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν κάθε φορά που βρίσκονται αντιμέτωποι με κάποια χημικά. Το τελευταίο θέμα που πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και που το θεωρώ προτεραιότητά μου είναι, όπως σας είπα, η προστασία των παιδιών από τις διαφημίσεις. Τα παιδιά εκτίθενται υπερβολικά ως καταναλωτές παρόλο που δεν καταναλώνουν με τον ίδιο τρόπο που καταναλώνουν οι ενήλικες, παρόλα αυτά επηρεάζονται από τις διαφημίσεις, άρα καταναλώνουν εντό αγωγικών διαφημίσεις. Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να κάνουν τους υπολογισμούς που πρέπει ή να αντιληφθούν τα πράγματα έτσι όπως οι μεγάλοι. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στη στρατηγική μας και να βρούμε έναν τρόπο για να προστατεύουμε τα παιδιά από τις διαφημίσεις. Τα παιδιά πρέπει να τα έχουμε πάντα υπόψη μας στις αποφάσεις μας και κυρίως εδώ στη νέα αυτή στρατηγική μας για τους καταναλωτές. Στόχος της στρατηγικής είναι να υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η ενημέρωση και η συνδυτοποίηση των καταναλωτών. Άρα να είναι εν γνώση τους όλοι οι κίνδυνοι και να μπορούν να αποφασίζουν εν γνώση των συνεπειών. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνετε ευκαιρία να συνεργαστώ με τους συναδέλφους για αυτό το θέμα. Σας έδωσα έτσι κάπως γρήγορα τις ε, προτεραιότητές μου και από εδώ και πέρα θα ακούσω με ιδιαίτερη προσοχή τους συναδέρφους. Ελπίζω όλοι μαζί να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε μια καλή στρατηγική προστασία των καταναλωτών και να επηρεάσουμε τα πράγματα έτσι όπως πιστεύουμε ότι πρέπει. Το 2012 ελπίζω οι παρατηρήσεις μας να λυθούν υπόψη. Δεν είναι αυτά όλα όσα είχα να πω, αλλά έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου. Εξάλλου είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων αυτή που κάνουμε. Θα επανέλθουμε. Περιμένω τώρα να ακούσω τους συναδέρφους. Και προσδοκώ στην εξαίρετη συνεργασία που είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε μεταξύ μας. Και αυτό γιατί είναι κοινό συμφέρον όλων μας να επηρεάσουμε την στρατηγική όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σβένσον, νομίζω έχουμε χρόνο να ακούσουμε και τους κοιόδης. Κυρία Γκριν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα και την κυρία Σβένσον που συνεννοήθηκε με τους σκιώδεις Η έκθεσή της μας δίνει την ευκαιρία να ξανασκεφτούμε το θέμα της καλύτερης δυνατής προστασίας των καταναλωτών και καταναλωτριών μέχρι το 2020. Και επειδή εδώ στην Επιτροπή μας επιμένουμε πάντα πολύ στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες και προτάσεις του Μισελ Μπαρνιέ, και θέλουμε όλο και περισσότερες και χρησιμότερες πληροφορίες για τους καταναλωτές και καταναλώτριες. Η έκθεση αυτή είναι πολύ χρήσιμη, υπήρχε και η έκθεση κάμπους προηγουμένως. Είναι φανερό λοιπόν ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ανησυχίες και ευχές των καταναλωτών αν θέλουμε να είναι χρήσιμη όντως αυτή η εσωτερική αγορά. Στο ΕΛΚ πιστεύουμε ότι ο κύριος στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής ως προς την προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών τα επόμενα χρόνια πρέπει να είναι η καλύτερη πληροφόρηση και η περισσότερη ευθύνη να είναι πιο πληροφορημένοι, να ξέρουν ακριβώς τι αγοράζουν και έτσι να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στην εσωτερική αγορά, σε μια δικαιότερη και σταθερότερη εσωτερική αγορά. Γι' αυτό νομίζω ότι η μελλοντική στρατηγική πρέπει να βασίζεται σε τρία πράγματα. Πρώτον, πληροφόρηση και των πολιτών και των καταναλωτών για τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους. Εξάλλου οι αριθμοί είναι εύγλωτοι για το ηλεκτρονικό ας πούμε εμπόριο ξέρουμε ότι είναι σημαντική μερίδα του γενικότερου εμπορίου και οι καταναλωτές διστάζουν πάρα πολύ να αγοράσουν ηλεκτρονικά. Μόνο 48% θεωρούν ότι έχουν εμπιστοσύνη να αγοράσουν ηλεκτρονικά και μόνο 33% όταν πρόκειται και για αγορά από ξένη χώρα ηλεκτρονικά. ενώ με τον παραδοσιακό τρόπο υπάρχει εμπιστοσύνη κατά 61%. Άρα ε, από τις δεύτερες μάλλον και τρίτες ηλεκτρονικές αγορές. Η πρώτη αγορά είναι η δύσκολη. Είναι λοιπόν σημαντικό να είναι καλύτερα πληροφορημένοι οι καταναλωτές και καταναλώτριες για τα προϊόντα που αγοράζουν, για τα δικαιώματα και τις ευθύνες τους ώστε να αγοράζουν πιο υπεύθυνα, πράγμα το οποίο σημαίνει βέβαια και ευθύνη των εμπόρων. Και εδώ φαίνεται από τους αριθμούς ότι οι έμποροι θεωρούν ότι γενικά γνωρίζουν την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, αλλά μόνο το 26% γνωρίζει σε ποια περίοδο μέχρι πότε μπορεί να επιστρέψει ένα ελαττωματικό προϊόν ο καταναλωτής. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Ως προς την γνώση ή άγνοια των εμπόρων για τις υποχρεώσεις τους. Γιατί πολλοί καταναλωτές έχουν γνωρίσει την περίπτωση όπου τους αρνείται ο έμπορος να επιστρέψουν το εμπόρευμα. Πρέπει λοιπόν να γίνει και μια καλύτερη αποτίμηση του κοινοτικού κεκτημένου. Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και καταναλωτριών ελπίζουμε να βελτιώσει τα πράγματα. Πολλά από αυτά που συζητήσαμε κατά την αναθεώρηση της οδηγίας ε, που συνίστανται σε καλύτερη εναρμόνιση και ελπίζουμε η εφαρμογή της από τα κράτη-μέλη να συνοδευτεί από καμπάνιες πληροφόρησης των καταναλωτών και καταναλωτριών και μέσω των οργανώσεών τους και μέσω των εθνικών αρχών. Όλα αυτά θα παίξουν ρόλο στην αποτίμηση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών και για τις πιθανές και ενδεχόμενες προσαρμογές που μπορεί να χρειαστούν και για τα φτηνά ταξίδια Όλα αυτά πρέπει να αποτιμηθούν, αξιολογηθούν και να δούμε μετά αν το κοινοτικό κεκτημένο λειτουργεί καλά και με τις καινούργιες τεχνολογίες. Άλλο στοιχείο τώρα, το οποίο θα το πούμε και αύριο, να διευκολυνθεί η πρόσβαση στις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης των διαφορών. Και τρίτον, η επιτήρηση των αγορών και της ασφαλείας των προϊόντων. Είναι και αυτό βασικό στοιχείο για την εμπιστοσύνη. Και εδώ οι αριθμοί είναι ενδιαφέροντες, μάλλον ενθαρρυντικοί αυτή τη φορά για την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά πρέπει να διευρυνθεί η προσπάθεια που γίνεται συντονισμού. Για τα ΑΠΕΞ είχαμε μιλήσει, είναι αποτελεσματικό εργαλείο για τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ χωρών μελών και οι σχέσεις μας με χώρες σαν την Κίνα ως προς την ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να ενισχυθούν και με αυτήν και με άλλες χώρες. Και τώρα τελειώνω κύριε Πρόεδρε, τελειώνω με μια λεξούλα για το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως είπα είναι τομέας με μεγάλο μέλλον όταν βέβαια αγοράζει κανείς κάτι από το ίντερνετ ιδίως όταν αφορά κάτι που μπορεί να επηρεάσει την υγεία του τρόφιμα και φάρμακα πρέπει να υπάρχει και τελωνιακός έλεγχος τέλος δεύτερο τέλος η πολιτική προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών σε επίπεδο κομισιών. Τουλάχιστον τρεις επίτροποι είναι αρμόδιοι για αυτό το θέμα. και που συνεργάζονται για να ανταποκριθούν σε αυτό το δύσκολο έργο που είναι όμως τόσο απαραίτητο για την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς. Θα ήθελα περισσότερη συνέπεια και συνοχή κάποιος επίτροπος από τους τρεις ας πούμε να είναι επισήμως ο συντονιστής και των τριών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ο κύριος ε, Ντάλι ε, μας είπε ότι έχει αυτή την αρμοδιότητα και ίσως και κάποιος μπορεί να το επιβεβαιώσει αργότερα. Η κυρία Γκέπχαρτ έχει τον λόγο και αν μείνει χρόνος θα μιλήσω κι εγώ. Εγώ θα είμαι λιγάκι πιο σύντομη. Θα ήθελα καταρχήν ε, να ζητήσω συγγνώμη από τον αδελφό μου ο οποίος ε, δεν μπορούσε να ήταν παρόν και μου έδωσε ένα σκιαγράφημα με τις ε, πρώτες του σκέψεις. Είναι έτσι απλά τροφή για συζήτηση, μια συζήτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους πολίτες, όπως και η κυρία Σβέντσεν. Και εδώ ευχαριστώ για την ε, πολύ καλή ε, ανακεφαλαίωση που έγινε. Η κυρία Σβέντσεν είπε ότι πράγματι στο επίκεντρο θα πρέπει να είναι τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτό είναι το α και το ω εκείνων που καλούμε να πράξουμε. Άρα δηλαδή σε όλες τις ε, προτάσεις που έχουν σημασία για τους καταναλωτές πρέπει να ξεκινάμε από τα δικαιώματα των καταναλωτών. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Βεβαίως ο συνάδελφος επισημαίνει ότι επειδή συνέχεια το θέμα του διαδικτύου. Επισημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν όλο και περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου, αλλά και εξίσου πολλοί που δεν το χρησιμοποιούν και δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ότι και σε αυτούς ε, πρέπει να προσφέρουμε υπηρεσίες κατάλληλες ε, στον τομέα της ε, πολιτικής για τον καταναλωτή να μην μιλάμε μόνο για διαδίκτυο, να μιλάμε και για όλα τα άλλα τα οποία πρέπει και να παραμείνουν. Και αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Τώρα, πληροφορίες για καταναλωτές και για επιχειρήσεις. Ενημέρωση. Αυτά είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να μπουν στο προσκήνιο και βεβαίως αυτά πρέπει να προσαρμόζονται στις ε, διάφορες ομάδες στόχο σε νέους, σε πιο ηλικιωμένου, σε άτομα με αναπηρία. Άρα δηλαδή να υπάρχει μια σειρά ε, επικοινωνίας ε, ανάλογα με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των καταναλωτών. Όχι δηλαδή μία και μόνο μέθοδος, αλλά μία σειρά ε, μεθόδων που θα προσαρμόζονται. Τέταρτο σημείο που θέλει να θίξει είναι το θέμα της έρευνας και στο δικό μας το πρόγραμμα πλαίσιο, αν το διαβάσει κανείς, δεν αναφέρεται ο καταναλωτής, παραλείπεται ο καταναλωτής. Αυτό λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε καλύτερη έρευνα για τις ανάγκες των καταναλωτών. Διότι κυρίως όσον αφορά την ε, πρόσβαση στις ε, πληροφορίες, όσον αφορά στις ε, μεθόδους ή ακόμα και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό και που το, το οποίο το έδειξε η κυρία Λεκρούπ, δηλαδή η εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων. Θα μιλήσουμε αύριο γι' αυτό και αυτό είναι ένα εξίσου σημαντικό θέμα. Πέμπτο σημείο που θα ήθελα να δείξει ο συνάδελφός μου είναι η εξή κατάσταση. Σε πάρα πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν ε, διάφοροι και διαφορετικοί φορείς ε, που είναι αρμόδιοι για το δίκαιο του καταναλωτή. Είναι λοιπόν απαραίτητο να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια έτσι ώστε οι καταναλωτές ε, να μπορούν να είναι καλύτερα ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και για τις υποχρεώσεις τους. Άλλα θέματα που θα ήθελε να θίξει ο συνάδελφος είναι παγκοσμιοποιημένη αγορά ε, σε σχέση με την επιτόπια αγορά Οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι μπροστά στην κατανάλωση, υπάρχουν πλούσιοι και λιγότερο πλούσιοι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, διαφορές ε, και στην παροχή των υπηρεσιών. Ε, υπηρεσίες ανατίθενται σε τρίτους. Με όλες τις συνέπειες. Καινοτομία. Καινοτομία της ε, τεχνολογίας ε, και των μέσων. Υπάρχει το θέμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Έχουμε μια όλο και μεγαλύτερη ομάδα πιο ηλικιωμένων πολιτών Και εδώ βέβαια αυτό που παίζει ρόλο είναι να υπάρχει συσχετισμός με πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, ε, την ενέργεια. Αυτά είναι λέξη κλειδί που σας αράβιασα. Λέξη κλειδί που μου τις είχε γράψει και εγώ τις διάβασα. Είμαι σίγουρη ότι αν ήταν εδώ θα είχε να πει πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά μπορώ να φανταστώ ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα να συζητήσουμε και εγώ ε, στηρίζω ανεπιφύλακτα όλα αυτά, τις, όλες τις λέξεις κλειδί που μου ε, έγραψε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και την εισηγήτρια που μας ε, περιέγραψε αυτό το σημαντικότατο θέμα. Η ανάλυση μας για μια στρατηγική προστασία των καταναλωτών και καταναλωτριών σε πολιετές πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πρώτα απ' όλα έναν απολογισμό. Πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο απολογισμός και ευχαριστώ την Κομισιόν που μας έδωσε πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα. Υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας που μας έδωσαν που όπως το λέμε εμείς working document και θέλω να πω κάτι γενικότερο συνεχώς θέλουμε περισσότερες πληροφορίες για προστασία του καταναλωτή και της καταναλώτριας και αυτό είναι θεμητό αλλά μπροστά μας έχουμε μια αγορά που συνεχώς καινοτομεί και στο μάρκετινγκ και στην τεχνολογία και τα κάνει τα πράγματα όλο και πιο πολύπλοκα. Δύο πολυπλοκότητες λοιπόν και άρα ο καταναλωτής και η καταναλώτρια μπορεί να μην χάνεται μεν εκεί μέσα αλλά δεν μπορεί να τα καταλάβει όλα και να οργανωθεί αναλόγως. Θέλω να καταλάβουμε εδώ ότι δεν αρκεί να λέμε ότι χρειάζεται περισσότερες και περισσότερες πληροφορίες για τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Γιατί όσο περισσότερες πληροφορίες του δίνουμε, όλο και πιο ακατάληπτες θα γίνονται για εκείνον. Εκτός αν έχει σπουδάσει καταναλωτής. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζουν οι συνάδελφοι ότι αφού γυράσκει ο πληθυσμός και είναι όλο και περισσότεροι οι θα ήταν καλό για το μέλλον να σκεφτούμε και κάτι και για αυτούς να έχουμε ορισμένους άξονες να ξέρουμε κάθε φορά για ποια στρατηγική πρόκειται παράδειγμα εγώ δεν τίθεμαι πολύ υπέρ της εφαρμογής ενός 28ου καθεστώτος όπως λέμε όπως λέει και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, όχι η ΝΟΜ, η ΝΟΜ, η Επιτροπή ΝΟΜ, ζουρί. Γιατί όλα αυτά θα δημιουργήσουν όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Γι' αυτό προτιμώ να ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο της εναρμόνισης. Είναι δύσκολο να υπάρξει μέγιστη εναρμόνιση, αλλά άμα δεν γίνει τελείως δεν είναι καθόλου χρήσιμη. Επίσης θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και καταναλώτριες και να μην ζητάμε τα πάντα. Το να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει μια επιλογή δεν σημαίνει να γνωρίζει απ' έξω ένα κάρο πληροφορίες αλλά πώς να διαχειριστεί την πληροφόρηση που διατίθεται. Αύριο το πρωί θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτά τα θέματα, αλλά πρέπει να βάλουμε υπόψη μας και τις οργανώσεις των καταναλωτών και καταναλωτριών και να μην λέμε πάντοτε να τις λάβουμε υπόψη, να τις λάβουμε υπόψη, αλλά να τις λάβουμε πραγματικά υπόψη. Έπειτα και τελειώνω εδώ. Είναι κάτι που προκύπτει σαφώς από τα έγγραφα της Κομισιόν. Η Ένωση αποτελείται από κράτη-μέλη που δεν έχουν ίδια μεταχείριση των καταναλωτών τους. Και πρέπει να υπάρξει εδώ προτεραιότητα τα επόμενα χρόνια που να συνίσταται στο ότι όλες οι χώρες της Ένωσης θα έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Να υπάρξει σύγκληση των συστημάτων, όχι απαραίτητο μέγιστη εναρμόνιση, αλλά τουλάχιστον να δοθεί ένα κίνητρο να ζητηθεί από τις χώρες μέλη να ακολουθήσουν αν έχουν λήψεις ε, άλλες χώρες να τα σκεφτούμε όλα αυτά στα πλαίσια αυτής της έκθεσης και να μην γίνει απλώς ένας κατάλογος όλων όσων πρέπει να γίνουν γιατί αυτά τα έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές για να προασπιστούμε τον καταναλωτή και την καταναλώτρια αλλά να σκεφτούμε πώς θα τα οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας κατευχαριστώ. Κοιτάξτε, έχουμε καθυστερήσει και ε, δεν θα μιλήσω. Ε, απλώς θέλω να πω ότι η προσέγγιση στον τηλεφώνη είναι η σωστή και θέλω να ενθαρρύνω όλους για το ότι από αυτή την έκθεση πράγματι μπορεί να προκύψει προσθέμενη αξία και πρέπει να μπούμε στη θέση του καταναλωτή. Η κυρία Σβέντσεν ανέφερε πολλά και κρίσιμα θέματα. Δεν είναι όλα αυτά στις δικές μας αρμοδιότητες, πρέπει όμως να τα σκεφτούμε. Και νομίζω όλη αυτή η ιδέα σχετικά με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των καταναλωτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η σκέψη πίσω από αυτή την πρόταση, όπως είπατε και αρκετοί από εσά, είναι ότι τώρα ε, καλούμεθα ε, να εξετάσουμε ε, νέα στοιχεία επειδή υπάρχει αυτό το νέο καθεστώς και πρέπει επίσης να σκεφτούμε και τα επιτεύγματα αυτής της νέας οδηγίας. Τώρα είναι μια καινούργια εκδοχή. Ε, υπάρχει η αναθεώρηση ήδη φυστάμενων οδηγιών, υπάρχουν και άλλες ε, νέες οδηγίες και νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι όλα αυτά να τα εξετάσουμε κάτω από το πρίσμα ε, των προσδοκιών του καταναλωτή. Η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται να υπάρχουν πολλές δημοθεσίες, απλά ε, να υπάρχει προστασία, να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα αν κάτι δεν πάει καλά. Βεβαίως εμείς εμπλεκόμεθα σε όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι ε, κυρίως στον Επίτροπο κύριο Ντάλι έχουμε πει ότι ε, εμείς τοποθετούμεθα έχοντας κατά νου ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Έχουμε την έρευνα ε, χαίρομαι που πάρα πολύ κοιτάνε αυτό το scoreboard του καταναλωτή, το βαθμολόγιο αν θέλετε. Υπάρχει μια βάση ανάλυσης. Ε, χαίρομαι που η κυρία Γκέπχαρτ μίλησε επίσης ε, για αυτό που αποκαλείται ορίζοντας 2020 το νέο ερευνητικό πρόγραμμα γιατί συμφωνώ μαζί της και το άλλο που θέλω να προσθέσω είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ρόλο της λιανικής πώληση. γιατί σε τελική ανάλυση ε, πού είναι το πρώτο σημείο επαφής ε, των ε, καταναλωτών. Είναι ο Λιανοπολιτής. Αυτός λοιπόν έχει την ευθύνη να εξετάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή. Βεβαίως έχει ευθύνη ο Λιανοπολιτής διαδικτυακά αλλά και ο απλός. Αυτό είναι το σημείο επαφής Αυτή ήταν η σύντομη παρέμβασή μου. Οι διερμηνείς μας έδωσαν πέντε λεπτά. Έχουμε εδώ δύο διευθυντές. Ένα λεπτό μπορείτε. Ο καθένας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Η κυρία Μάινο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι αρκετοί συναδελφοί σας αναφέρθηκαν στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας, όπου απαιτείται ε, η πολιτική του καταναλωτή ε, να ενταχθεί σε όλες τις πολιτικές της Επιτροπής. Και από εκεί προέκυψε η οδηγία με την οποία θέλουμε ένα όραμα το οποίο θα ε, συμπεριλαμβάνει σε ένα και μόνο έγγραφο οτιδήποτε προτίθεται να κάνει η Κομισιόν για να ε, προάγει τα δικαιώματα, την ασφάλεια, τη θέση του καταναλωτή στην ε, κοινή αγορά. Οι προκλήσεις που εντοπίσατε εσείς είναι αυτές που εντοπίσαμε και εμείς, όλο και μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, ψηφιοποίηση, και γύρανση πληθυσμού. Αυτό αποτελεί τόσο ευκαιρία αλλά δημιουργεί και προκλήσεις. Ε, διάρκεια πρέπει να συνεργαστούμε επ' αυτού ε, με τους ε, συναντέλφους μας από το περιβάλλον. Πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Η Γενική Διέτη ΣΑΝΚΟ αναφέρεται στο ότι πρέπει να περιορίσουμε τα τρόφιμα που πετιόνται. Ασφάλεια όλες οι φορεί, όλοι οι φορείς, οι οργανισμοί θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των κατοίκων τους. Ε, Ράπεξ ε, συνεργαζόμαστε και με ε, συνεργάτες μας σε τρίτες χώρες, όπως είπε ο κύριος Ρος, ο καταναλωτής χρειάζεται να αισθάνεται ότι συμμετέχει και αυτός στην κοινή αγορά της Ευρώπης. Οι απαιτήσει του καταναλωτή πρέπει να εισακούνται τόσο δυνατά όσο και οι απαιτήσει της βιομηχανίας. Ε, το αν πρέπει να περιορίσουμε τις πληροφορίες που δίνονται στον καταναλωτή. Εκεί ίσως ε, έχουμε ε, ενδιάμεσους ε, που αφορούν και τους λιανοπολιτές και αυτοί πρέπει να εκπαιδευτούν για τις υποχρεώσεις τους που σε γενικές γραμμές όμως είναι πολύ πρόθυμοι. Και το τελευταίο που θέλω να αναφέρω είναι να συντάξει ένα έγγραφο και τα δικαιώματα επίσης είναι σημαντικό αλλά θα πρέπει να γίνονται ε, πραγματικότητα με τη σωστή εφαρμογή. Αυτό λοιπόν που προτείνει ο κύριος Τάλι είναι μια ε, εναλλακτική ε, μορφή διαθέτησης διαφόρων, διαφορετικές αποζημιώσεις και θα κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά το δίκτυο προστασίας καταναλωτή το οποίο βοηθάει σε διασυνοριακό επίπεδο. Εγώ θα μιλήσω λιγότερο. Τώρα θα μιλήσω λιγότερο από ένα λεπτό. Θέλω απλώς να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναήρθα μετά από τις ημερίδες για τα δικαιώματα των καταναλωτών και καταναλωτριών. Συνεργαζόμαστε η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ και ο Επίτροπος Ντάλι για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές από το Φεβρουάριο του 12. Εκτιμήσαμε ιδιαίτερα όλα όσα είπατε σήμερα και ένα μόνο έχω να προσθέσω ότι πολλά έχουν ήδη γίνει. Πρέπει τώρα να αποδειχθεί ότι είναι χρήσιμα με, τη με το νέο πρόγραμμα των καταναλωτών και επίσης να βρούμε μια εξισορρόπηση στην πρωτοβουλία αυτή. Έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη τα επόμενα χρόνια στην Επιτροπή μας πρέπει να αναθεωρήσουμε, την Επιτροπή σας, πρέπει να αναθεωρήσουμε, στην ε, τωρινή σύνθεση μάλλον της Κομισιόν, πρέπει να αναθεωρήσουμε τα πράγματα και τελικά να καταλήξουμε στο να βάλουμε τον καταναλωτή και την καταναλώτρια στη βάση κάθε πολιτικής έτσι ώστε το σύστημα να δουλεύει από την αρχή μέχρι το τέλος για να είναι πραγματικά τα δικαιώματά τους. προσμένο στη συνέχεια και χαίρομαι ιδιαίτερα για την καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σβένσον, φοβάμαι ότι τελείωσε ο χρόνος. Να σας δώσω μόνο το χρονοδιάγραμμα. Δεν έχετε την ευκαιρία να καταλήξετε άλλη φορά. Λοιπόν, στις 19 Σεπτεμβρίου θα εξετάσουμε την εκθεσή σας. 22 λίγη διορία κατάθεσης τροπολογιών και τον Οκτώβριο στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους διερμηνείς που μας έδωσαν αυτό το ζωτικό δεκάλεπτο παραπάνω. Θα ξαναβρεθούμε αύριο το πρωί εδώ. Λίγη